morning everybody, welcome. Um, Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ γεμάτη μερσιά διάταξη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση, καταρχάς της μερσιάς Έχω να προτείνω κάποιες τροποποιήσεις μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για το μέσο εμπορικής άμυνας, το μηχανισμό εμπορικής άμυνας, το Ολομέλεια, με εσύ τον κύριο Φιέλνερ, θα πρέπει να αποφασίσουμε τη διαπραγματευτική εντολή με το Συμβούλιο. Αυτό θα το συζητήσουμε υπό το σημείο 17α. Εντολή διαπραγμάτευσης. και θα αποφασίσουμε για την αντιπροσωπεία. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Ο συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο, μας ακούει ο κόσμος δηλαδή, η συνεδρίασή μας. Υπάρχει ο κατάλληλος αλληλογραφια Χθε συνεδρίασε η Διευθύνουσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΑΠΟΕ κατόπιν πρωτοβουλία στο κοινοβουλίο μας και των Κοινοβουλίων της Δικοινοβουλευτικής Ένωσης. Αποφάσισα λοιπόν να καλέσουμε τους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να παραστούν στην συνεδρίασή μας. συμπρόεδρος της Διακοινοβουλευτική ε, Επιτροπής και συγκεκριμένα αυτής της Διευθύνουσας Επιτροπής είναι ο κύριος Έρν Γέντερ, τον οποίο καλό να έλθει στο βήμα και βλέπετε ότι είναι ήδη εδώ. Χθε εγκρίναμε ένα ψήφισμα στο τέλος της συνεδρίασης το οποίο μπορείτε να βρείτε εκτός της αίθουσας αν σας ενδιαφέρει. πρόσφατα εμπορικά νέα έτσι ένα απάνθισμα Πρόοδος ε, στις διαπραγματεύσεις ε, ΕΠΑ, οικονομική συνεργασία δηλαδή με την ΕΚΟΑ στη Δυτική Αφρική. Έχουμε καταλήξει συμφωνία. Δεύτερον, υπάρχει και μια ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων για πολυμερείς ε, συμφωνίες ε, για τα περιβαλλοντικά καθώς στο πλαίσιο του ΠΟΕ. και με μη προτιμησιακή βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, Κίνα, και η Ιαπωνία θα συμμετάχουν στις δραματεύσεις αυτές. Πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Περνάμε στο σημείο 3. Το χρεωτικό θέμα, δυνάμει του κανονισμού δηλαδή, πρέπει να το συστήσουμε οπωσδήποτε στην Επιτροπή μας και πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσουμε αν θα κρίνουμε αυτή τη ε, συμφωνία του Συμβουλίου σε σχέση με έναν ε, κανονισμό, μάλλον διαδικασίες εφαρμογής για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ε, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σερβίας και προσωρινή συμφωνίας με τη Σερβία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πάνω να αποδεχόμαστε τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Για να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια πριν λήξει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδο, ή το αργότερο τον Απρίλιο. Προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών 6 το απόγευμα σήμερα, ακριβώ, 6 ώρα ακριβώ σήμερα για να ψηφίσουμε αύριο. Ο Ιούλιο Βίνκλερ που ήταν και εισηγητής στην πρώτη ανάγνωση είναι εισηγητής και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει εισηγητής και για τη δεύτερη ανάγνωση. Θα σας δώσω λοιπόν κύριε συνάδελφε το λόγο για να μας μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Λάβαμε τη θέση του Συμβουλίου για τον κανονισμό εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία. Ένας πιο παλιός φάκελος, το γνωρίζετε καλά αγαπητοί συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση με βάση την έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ τον Οκτώβριο του 2012 ένα θέμα το οποίο είχε σχέση και με το Trade Omnibus 1 αλλά ε, σταμάτησαν οι διαπραγματεύσει λόγω της διασύνδεσης ε, για ένα χρόνο τουλάχιστον με το Συμβούλιο. Ε, το Νοέμβριο επιτέλου πέρυσι επετέφθη η συμφωνία η οποία αντικατοπτρίζει και την έκφαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Omnibus 1 και επίσης το ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση με τη Σερβία. Η θέση του Συμβουλίου, όπως ε, έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή μας, ε, ε, βρίσκει, την χάνει τη Συμφωνία Δυνάμεις. Βέβαια υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, επιτυγχάνει την συνέπεια και συνεκτικότητα με τον κανονισμό που είχε τροποποιηθεί με την εμπορική δέσμη Omnibus 1 και δεύτερον με την πρόταση πάβουν οι αναφορέ πλέον στην προσωρινή συμφωνία, στην διάμεση συμφωνία. Έτσι έπρεπε άλλωστε να γίνει. Είναι Πολύ σημαντικό ο κανονισμό αυτό να τεθεί σε ισχύ χωρί άλλη καθυστέρηση, ώστε οι εμπορικές διατάξεις της συμφωνίας ε, σύνδεσης να μπορέσουν να ε, ισχύσουν προ όφελο των οικονομικών φορέων. Προτείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε να εγκρίνουμε τη θέση του Συμβουλίου χωρί τροπολογίε, διότι αντικατοπτρίζει τη δική μα θέση και ελπίζω και οι διακεκριμένοι συνάδελφοι να στηρίζουν στηρίξουν στην Επιτροπή αυτή το σχέδιο συστάσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Έχετε το σχέδιο συστάσεων στους φακέλους σας. Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξουμε τον εισήγητή μας αύριο στην ώρα της ψηφοφορίας. Ας κάνουμε τώρα όμως μια μικρή διακοπή για να σας πω ότι έχουμε και τον κύριο Σβέντεφερ που θα έρθει. Ε, δεν έχει έρθει όμως ακόμη, σε δύο-τρία λεπτά. Ο κύριος Αζεβέδο, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Uh, uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά να σας παρουσιάσω κάποιον βέβαια που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο κύριος Ρομπέρτα Ζεβέδο είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και είναι κατάλληλη χρονική στιγμή, επίκαιρη, έρχεται εδώ να μιλήσει σε εμάς. Νομίζω το Σεπτέμβριο λάβετε τα καθήκοντα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έρχεται εδώ, όταν έλαβε τα καθήκοντά του. Είχαμε και τα πρόσφατα επιτεύγματα του ΠΟΕ, από ε, την ηγεσία του με την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Παλί. Όσοι από εσά ήσασταν στον Παλί, πήγε την προσωπία του Κοινοβουλίου με κεφαλή στον υποφαινόμενο στον Παλί. και για όσους δεν έζησαν αυτές τις πολύ έντονες ημέρες στον Παλί, ε, θα σας πω ότι εμείς που ήμασταν εκεί θα, μπορέσω να το, θα το διατυπώσω όσο να τον πιο ε, μετροπαθώς μπορώ. Είδαμε τις εξαιρετικές ε, διαπραγματευτικές ε, ικανότητες του νέου Γενικού Διευθυντή για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. το κοινοβούλιο μας και αυτή η Επιτροπή πάντα λέμε ότι στηρίζουμε τον ΠΟΕ και το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε αυτούς τους διμερείς κανόνες και χαίρομαστε πολύ που η πρώτη συμφωνία που επετεύχθη μετά το γύρο της Ντόχας. Είναι βέβαια ίσως ένα μικρό κομμάτι στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα, αλλά εξακολουθεί να σημαίνει αναζωγόνηση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Τώρα βέβαια πρέπει να υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή. Έχουμε το, το Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και πολλά άλλα θέματα θα δούμε και τα επόμενα βήματα, τα επόμενα στάδια, αλλά ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ξανά σε τροχιά ο γέρος της Ντόχα. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Γενική Διευθυντά που ήσασταν εδώ. Χθες, όπως έλεγα νωρίτερα, και κατά σύμπτωση ε, συνεδρίασε η Διευθύνουσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης ε, του ΠΟΕ. Την κοινή αυτή ε, πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, την παρουσία σας συνοδέλφους ε, είπα ότι εγκρίναμε και ένα ψήφισμα. Το έχω μαζί μου εδώ και σας δίνω και το πρώτο αντίγραφο. Με πολύ μεγάλη χαρά. <coughs> Βρίσκεται εδώ και ο συμπρόεδρος της Διευθύνωσης Επιτροπής από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, ο κύριος Έρν Φιέντερ. Κάθεται και αυτός εδώ στο βήμα. και αυτό προς εκτίμηση της ε, ε, καλή συνεργασία που έχουμε στο πλαίσιο αυτής της ε, Διευθύνουσης Επιτροπής. Είναι πρώτη φορά που παρίστατο συμπρόεδρος από την Δικοινοβουλευτική Ένωση. Θα σας ακούσουμε λοιπόν κύριε Γενική Διευθυντά, μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τα μέλη της Επιτροπής και επίσης θα παρακαλέσω και τα άλλα μέλη της Διευθύνουσης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης των ΠΟΕ να λάβουν το λόγο εφόσον το επιθυμούν. Παρακαλώ κύριε Αζεβέδο, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλες και όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά χαρά για μένα που βρίσκομαι παρόν εδώ. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε να σας ομιλήσω σήμερα και ιδίως ευχαριστώ τον καθηγητή Βιτάλ Μορέιρα, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, καθώς και τον κύριο Όρν Φιέντερ, που είναι ο επικεφαλής της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και, την, και το ψήφισμά σας, θα το διαβάσω προσεκτικά, να είστε βέβαιοι. Και σίγουρα διότι το έργο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΠΟΕ είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του πολυμερού συστήματος. Ως βουλευτές όχι μόνο κυρώνεται και εγκρίνεται τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γενέβη και τα εξηγείτε και στο κοινό των χωρών σας, αλλά συνδέεται και τον ΠΟΕ ως οργάνωση με τους ανθρώπους τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει, δηλαδή τους πιο φόρου σας. Βασιζόμαστε σε εσά μέσω των κυβερνήσεών σας αλλά και μέσω φόρουμ όπως το παρόν να διαβιβάσετε τις ανησυχίες των ανθρώπων στις ε, κοινότητές σας. Είναι πολύ σημαντικός ο σύνδεσμος αυτός για να εξασφαλίσει ότι το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου θα λειτουργήσει και στο τοπικό επίπεδο. Δεν θέλουμε στη Γενέβη να είμαστε μια απομονωμένη νησίδα. Θέλουμε να λειτουργούμε με προσκλάθα κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει στενές και ισχυρές ε, σχέσεις με τους βουλευτές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μιας και είναι η πρώτη μας ε, συνάντηση μετά το Μπαλί, με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω για πρώτη φορά για την επιτυχία της υπουργική Διασκέψεως. Ορισμένοι από εσά ήσασταν μάλιστα και παρόντες ή παρούσες. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να συναντηθούμε διότι είχα βέβαια αρκετά πράγματα να προλάβω. Με την ευκαιρία όμως σήμερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την η υποστήριξη που προσφέρατε και στον πάλι στις προσπάθειες που έχουμε αναλάβει όλοι για να καταλήξει ο ΠΟΕ στην πρώτη του διεθνή πολυμερή συμφωνία από το 1995 όπου ιδρύθηκε. Σίγουρα το Παλί ήταν ιστορική στιγμή για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Απέφερε σημαντικά κέρδη για την παγκόσμια οικονομία και για τις αναπτυγμένες και για τις αναπτυσσόμενες και για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το πακέτο του Μπαλί θα προσφέρει σημαντική όθηση στην παγκόσμια οικονομία με δημιουργία απασχόληση και ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα. Όμως το Μπαλή ήταν ιστορικό και διότι για πρώτη φορά απέδειξε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα μετά από πολυμερή διαπραγμάτευση. Είναι σημαντικό διότι ξεκινά μια νέα εποχή για το ε, πολυμερές εμπορικό σύστημα και για τον ίδιο τον ΠΟΕ. Βέβαια, το Μπαλί δεν ήταν το τέλος, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Αντίθετα, είναι η αρχή της διαδρομής. Είμαστε ακόμα μακριά από την ολοκλήρωση του έργου μας. Έχουμε δε μπροστά μας δύο σημαντικά ε, καθήκοντα. Και το πρώτο είναι βέβαια η εφαρμογή των αποφάσεων του Μπαλί. Οτιδήποτε θα κάνουμε από εδώ και μπρος θα αποδεικνύει ή δεν θα αποδεικνύει την αξιοπιστία μας ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι βέβαια ότι η διακήρυξη του Μπαλί καλεί τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να καταστρώσουν ένα σαφώς ορισμένο πρόγραμμα εργασιών για τα υπολοιπόμενα θέματα της ατζέντα ανάπτυξης της Ντόχα και αυτό μέχρι το τέλος του 2014. Έτσι λοιπόν η πραγματική σκληρή δουλειά τώρα αρχίζει. Τα δύο αυτά καθήκοντα θα αποτελέσουν βέβαια και τον κύριο όγκο της εργασίας μας, των εργασιών μας για, τα, για το υπόλοιπο του έτους. Και αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν στην ομιλία μου σήμερα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την εφαρμογή. Όπως είπα και πριν λίγο, η πραγματική σημασία του πακέτου ή της δέσμης του Μπαλί και της υλοποίηση των στόχων είναι ότι θα επιτευθούν μόνο μετά από την ολοκλήρωση των δράσεων που θα αναλάβουν τα μέλη του ΠΟΕ τους επόμενους μήνες. Και αυτό είναι σημαντική δοκιμασία για το σύστημα και πρέπει να την περάσει η δοκιμασία αυτή αν θέλουμε να ε, υλοποιηθούν τα αγαθά αποτελέσματα του Μπαλί. Αυτή η πρόκληση λοιπόν είναι πολύ σημαντική, ιδίω για παράδειγμα στην Συμφωνία για την Διευκόλυνση του Εμπορίου, δοθέντος του, εύρου, του εύρους και της περιπλοκότητας της Συμφωνίας, καθώς και του μεγέθους των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Η απόφαση που λάβαμε να πλουστεύσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις διαδικασίες τελωνίων, να τις κάνουμε πιο διαφανείς και να μειώσουμε το κόστος των συναλλαγών, περιλαμβάνουν και ορισμένα στοιχεία και ιδίω την παροχή τεχνικής στήριξης για την υποστήριξη αναπτυσσομένων και λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις και να μπορέσουν έτσι να συμμετάσχουν στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Έχουμε αρχίσει τη δουλειά λοιπόν ήδη στη Γενέβη προς την κατεύθυνση αυτή για να εξασφαλίσουμε την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Διευκολύνσεως του Εμπορίου με την πρώτη συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου πρόεδρος εκλέχθηκε ο πρέσβης Εστεμπάν από τις Φιλιππίνες. Η επιτροπή που ανέφερα, η προπαρασκευαστική επιτροπή, θα αρχίσει λοιπόν σύντομα να εκπονεί σχέδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που έλαβε από τους υπουργούς στον Παλί και ιδίως για να εξασφαλίσει την θέση σε εφαρμογή της Συμφωνίας του Εμπορίου. Θα χρειαστούμε την βοήθειά σας ως βουλευτών για να εξασφαλίσουμε ότι η Συμφωνία θα ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδικασία κυρώσεων έτσι ώστε να μπορέσει έγκαιρα να τεθεί σε ισχύ. Η ικανότητά μα όμω να προχωρήσουμε ολόκληρη την ατζέντα του ΠΟΕ προ τα Εμπρό, εξαρτάται από την ικανότητά μα πάλι να εκπληρώσουμε τι δεσμεύσει για την παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Για να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές η Γραμματεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα αξιολόγησης αναγκών για να εντοπίσει τι είδους στήριξη θα χρειαστούν οι χώρες αυτές και μάλιστα να γίνει αυτό το δυνατόν συντομότερο. Οι κράτη δωρητές αλλά και διάφορες οργανώσεις δωρητών επίσης ετοιμάζονται να προσφέρουν την ζωτική υποστήριξη στην διευκόλυνση εμπορίου. Προεβδομάδος συναντήθηκα με τους προσώπους 25 χωρών και οργανώσεων για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την σημασία της συνεργασίας για την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου βεβαίως θα συμβάλλει στην διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ δωρητών και ε, απολυπτών ή δικαιούχων. Και εκεί θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο οι βουλευτές. Βέβαια, η διευκόλυνση εμπορίου δεν ήταν παρά ένα μόνο στοιχείο της δέσμης του Μπαλί, διότι εκεί δέκα αποφάσεις ελήφθηκαν συνολικά, από τις οποίες τέσσερις για την γεωργία, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ε, ατζέντα ανάπτυξης της ΔΟΧΑ... που απασχολεί τον ΠΟΕ ήδη από το 2001. Ήταν λοιπόν σημαντικό να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός στην γεωργία, όμως τα μέλη μας ήταν ρεαλιστές για το πώς θα γίνει αυτό. Ήταν σαφές ότι έδειξε προθυμία η Ευρώπη να συμβάλλει στην γεωργία και αυτό βεβαίω αναλογικά με το τι θα γίνει σε άλλου τομεί τη διευκόλυνση εμπορίου. Πράγματι πρόκειται για ένα ρεαλισμό, τον οποίο εκτίμησαν νομίζω τα άλλα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έγιναν λοιπόν σημαντικά βήματα στον Παλί, για παράδειγμα για τι επιδοτήσει εξαγωγών και άλλα μέτρα με παρόμοια αποτελέσματα και επιτεύχθηκε και πρόοδο για την εφαρμογή των ποσοστώσεων στις ε, υποχρεώσεις που έχουν αληφθεί ήδη από τον γύρο της Ουρουάης. Και έγινε και μια επανεπιβεβαίωση των πολιτικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Χονγκ Κονγκ για το Βαμβάκι, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλές αφρικανικές χώρες. Η δέσμη προβλέπει επίσης να γίνουν διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προμηθειών τροφίμων και θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ε, σιτηρών για να διανεμηθούν μετά στους φτωχότερους. Λήφθηκαν αποφάσεις και για θέματα ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ένα ειδικό πακέτο για τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες που ήταν πραγματικά επιτυχία κλειδί της Υπουργικής Διάσκεψης του Μπαλί και σημαίνει και είναι ένα μάλλον ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη ένταξη των ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών στο πολυμερές εμπορικό σύστημα. Μεταξύ αυτών, μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν να αποκτήσουν νέες εξαγωγικές ευκαιρίες οι ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες. Βελτιώσεις σε συστήματα προτιμήσεων που επεκτείνουν τις εξαιρέσεις από δασμούς και ποσοστώσεις στις εξαγωγές των ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών. Επίσης υπήρξε μια συμφωνία για την απλούστευση των κανόνων προέλευσης που συνοδεύουν συνήθως τα ανοίγματα αυτά και που θα επιτρέψουν την βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης στις αγορές των ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών. Και εδώ πάντως το μπαλί δεν σημαίνει παρά μόνο την αρχή. Δεν είναι το τέλος. Χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά να γίνει για να μετατραπούν οι αποφάσεις αυτές και ιδίω οι ε, αποφάσεις που θα ωφελήσουν τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες σε πραγματικά κέρδη. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή με ιδιαίτερη στόχευση από όλα τα μέλη στις πρωτοβουλίες αυτές. Τώρα ευρύτερα και κάτι που αφορά όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες, υπήρξε η απόφαση να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης που να επιτρέπει την εξέταση και ενίσχυση ειδικών διατάξεων προτιμησιακής μεταχείρισης. Αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης θα επιτρέπει λοιπόν να εξετάζεται αν έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιούνται οι προτιμήσεις αυτές και να προτείνει και βελτιώσεις. Όλες αυτές οι δέκα αποφάσεις λοιπόν σημαίνουν μια πραγματική πρόοδο. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ εργάστηκαν σκληρά πέρσι για να μπορέσουν να οδηγήσουν σε αίσιο πέρας το πακέτο του Μπαλί. Η δική μου αίσθηση τώρα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο αυτό για να καταλήξουμε στα ευεργετικά αποτελέσματα του πακέτου. Και γι' αυτό ζητώ και πάλι την υποστήριξή σας για να διατηρήσουμε την ορμή, την όθηση που επιτύχαμε στο Μπαλί. Όπως είπα, η εφαρμογή της συμφωνίας είναι το πρώτο βήμα, ο πρώτος στόχος μας. Το δεύτερο είναι να αρχίσουν, να επαναληφθούν μάλλον οι συνομιλίες και να οριστεί ξεκάθαρα ένα πρόγραμμα εργασιών για τα υπόλοιπα θέματα της Ατζέντα ε, Ανάπτυξης Ντόχα μέχρι το τέλος του 2014. Έχω ακούσει προσεκτικά τα όσα μου είπαν τα μέλη σχετικά με το πώς θα πρέπει να το επιτύχουμε αυτό και νομίζω ένα πράγμα έχει προκύψει ξεκάθαρα. Για να μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα και προς τα πίσω και να μάθουμε από τα σφάλματα του παρελθόντος διότι αρκετά έγιναν αλλά έχουμε τώρα και μια ιστορία επιτυχίας, τον Παλί. Ας διδαχθούμε λοιπόν και από αυτό. Ας διδαχθούμε και από τα σφάλματα του παρελθόντος αλλά και από τις επιτυχίες. Το Παλί μας πρόσφερε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό καλών διδαγμάτων για το πώς μπορούμε να είμαστε επιτυχείς πολυμερός. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο να επαναλάβουμε την προσέγγιση που επιτύχαμε για τον Παλίο, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα δύσκολα θέματα και μπορέσαμε έτσι να επιτύχουμε ε, σημαντικές πρόοδους σε περιφερειακά θέματα, αν και βέβαια η διευκόλυνση εμπορίου δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι περιφερειακό θέμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας μέχρι τώρα έχουν τονίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολυμερής συμφωνία θα απαιτήσει κάποια αποτελέσματα ειδικά στον τομέα της γεωργίας. Και εφόσον η γεωργία μπει στις συζητήσεις αυτής, αυτές, τα δύο άλλα σκέλη του τρίποδα αυτού θα παίξουν και αυτά. Δηλαδή τα βιομηχανικά αγαθά και οι υπηρεσίες. Γνωρίζω βέβαια ότι αυτή είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υφίσταται αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ των τριών ε, σκελών. Για να συζητήσουμε όμως συλλογικά τα, τα, τα ζητήματα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε και τις ευαισθησίες που ε, είναι αναπόσπαστο μέρος όλων αυτών των θεμάτων. Η Γεωργία για παράδειγμα θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί πολύ προσεκτικά δεν επιθυμώ να επαναλάβουμε ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν, διότι οι προσπάθειες εκείνες δεν αποδείχθηκαν επιτυχείς όπως το γνωρίζετε. Αναζητώντας όμως νέες προσεγγίσεις θα χρειαστεί μια πραγματική αξιολόγηση, μια πραγματική εκτίμηση των ευαισθησιών που υπάρχουν και βεβαίως και εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να στοχεύσουμε βεβαίως σε, κάποιες, σε κάποια σκόπιμες εκβάσεις, σκόπιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη και τους πολιτικούς περιορισμούς για κάθε θέμα σε κάθε χώρα. Πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί μια ισορροπία σε όλους τους τομείς διαπραγματεύσεων, όχι μόνο επομένως στη γεωργία, αλλά και στα βιομηχανικά αγαθά και στις υπηρεσίες. Αν δεν το κάνουμε αυτά, φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να επαναλάβουμε τον παλί ακριβώς, ωστόσο υπάρχουν διδάγματα που προκύπτουν από αυτό που πρέπει να διατηρούμε να έχουμε 200 υπόψη μας. Και μιλώντας με τα μέλη, αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένε ορισμένες παράμετροι ήδη έχουν ανακύψει και αποτελούν το πλαίσιο τη συζήτηση αυτή. Θα μιλήσω για ορισμένες από τις παραμέτρου αυτές τώρα, όπως τις αντιλαμβάνομαι εγώ, παρόλο που τονίζω ότι δεν πρόκειται για εξαντλητικό κατάλογο των παραμέτρων που θα σα αναφέρω, ούτε τι έχω βάλει με κάποια σειρά σημασία ή προτεραιότητα. Ο στόχος είναι μοναχά να προσφέρουν κάποια έμπνευση για τις συζητήσεις που θα διεξαγάγουμε. Πρώτη λοιπόν παράμετρος είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη πρέπει να διατηρηθεί ως ο κεντρικός πυλώνας των προσπαθειών μας. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε απτά αποτελέσματα υπέρ των φτωχότερων μελών. Δεύτερο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να στοχεύσουμε στα πράγματα εκείνα τα οποία είναι και εφικτά αντί να επιδιώκουμε αφηρημένους στόχους, ας εξετάσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε στόχους που να είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ φιλοδοξιών και ρεαλισμού. Η τρίτη παράμετρος είναι ότι τα μεγάλα θέματα της ε, Agenda Doha διασυνδέονται και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα μαζί. Και πάλι λοιπόν, το Μπαλί, όπως αποδείχθηκε και στον Παλί, το κλειδί είναι η ισορροπία. Πρέπει να βρούμε μια προσέγγιση στην οποία να συμβάλλουν όλα τα μέλη και από την οποία να υποφελούνται όλα τα μέλη. Το πάλι πέτυχε διότι όλα τα μέλη ήθελαν και κανένας δεν αντιμετώπισε αδύνατες να υλοποιηθούν απαιτήσει. Το τέταρτο είναι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ότι πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να έχουμε ανοιχτό μυαλό απέναντι σε νέες ιδέες που ίσως επιτρέψουν στα μέλη να αντιμετωπίσουν τα πιο δύσκολα εμπόδια. Η δημιουργικότητα αυτή ωστόσο πρέπει να συμβαδίζει και με την εντολή της ατζέντα της Ντόχα που όμως είναι αρκετά εύκαμπτη ώστε να επιτρέπει και νέες οδούς. Πέμπτο, η διαδικασία θα πρέπει να συνεχίσει να είναι τέτοια που να συμπεριλαμβάνει όλους, να είναι διαφανής και να συμμετέχουν σε αυτήν όλα τα μέλη σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο Μπαλί. Αυτό βέβαια κάνει πιο αργές διαπραγματεύσεις, αλλά παρόλα αυτά πετύχαμε. Μπορεί ορισμένε αντιπροσωπείε να προτιμούσαν κάποιε διαφορετικέ διατυπώσεις στη συμφωνία τελικά. Γνώριζαν όμω για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένε διατυπώσει. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την τελική αποδοχή του πακέτου. Έκτον, οι προσπάθειες μας θα πρέπει να γίνουν και μια αίσθηση του επίγοντος. Και αυτό ήταν σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του Μπαλί και δεν μπορούμε να περιμένουμε ξανά 18 χρόνια μέχρι ότου υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο να είμαστε προσεκτικοί, να μην βιαστούμε υπερβολικά και πέσουμε σε άλλο κύκλο αποτυχιών λόγω κακού σχεδιασμού. Τέλος, νομίζω επίσης ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα απέναντι σε νέες ιδέες όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις που θα λάβουμε μαζί, αλλά και σε ό,τι αφορά το εύρος των επόμενων βημάτων. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι το άλμα που ε, θα κάνουμε την επόμενη φορά. Όλα διαμιάς ή θα προχωρήσουμε με μικρότερα βήματα. Βεβαίως αυτό που θα προτιμούσαμε θα ήταν να ολοκληρωθεί ο γύρος και δυνατόν αμέσως. Ίσως να μπορέσει να γίνει σε ένα βήμα, ίσως να χρειαστούν περισσότερα βήματα. Πάλι αυτό θα είναι, όπως σας είπα, κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Και η συζήτηση αυτή έχει ήδη αρχίσει. Εγώ απίθυνα το λόγο στην Επιτροπή Διαπραγματεύσεων Εμπορίου στον ΠΟΕ την προηγούμενη εβδομάδα με παραπάνω από 30 εκπροσώπους οι οποίοι έλαβαν τον λόγο, αντιπροσωπείες δηλαδή, και με ικανοποίησε πολύ η θετική και επικοδομητική νότα που χρησιμοποίησαν στις ομιλίες τους. Τις επόμενες εβδομάδες θα συναντηθώ και με τους επικεφαλείς των διαπραγματευτικών ομάδων για να συζητήσω θέματα μαζί τους στην βάση των παραμέτρων που σας ανέπτυξα. Βέβαια, ένα άλλο θέμα για την ε, trade agenda είναι και άλλες πρωτοβουλίες εμπορίου, είτε πρόκειται για πολυμερείς, περιφερειακές ή και διμερείς Αυτές γίνονται ταυτόχρονα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως εμπλέκεται σε έναν αριθμό τέτοιων πρωτοβουλειών. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει έναν αριθμό διμερών συμφωνιών, έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις Ενωμένες Πολιτείες για την TTIP, έχει συμμετάσχει σε πολυμερείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία για τις Υπηρεσίες καθώς και για την ε, τεχνολογία της πληροφορικής. Έχω λοιπόν να πω κάτι και γι' αυτό. Όπως είπα και πριν, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι θετικές και καλοδεχούμενες, αλλά δεν μπορούν παρά να αποτελούν ένα μέρος μόνο της συνολικής εικόνας. Συμφωνίες όπως αυτές δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν κέρδη στο παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, ο πολλαπλασιασμός ρυθμίσεων και προτύπων προκαλούν περισσότερα κόστη αντί να τα μειώνουν. Όπως γνωρίζετε, το πολυμερές εμπορικό σύστημα ποτέ δεν είχε τον σκοπό να είναι η μοναδική επιλογή για τις διεθνείς εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις. Ήταν ένα σύστημα το οποίο συνυπήρχε με άλλες πρωτοβουλίες, χωρίς το ένα να αποκλείει το άλλο. Εν τέλει, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια τέτοια πρωτοβουλία και σαφώς είναι μια η οποία προωθεί και στηρίζει το πολυμερές σύστημα. Και είναι πραγματικό ότι οι διάφοροι κλάδοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου πρέπει να αναπτυχθούν για να μειωθεί το κενό μεταξύ των πολυμερών συμφωνιών και της νέας γενιάς συμφωνιών που διαπραγματεύονται εκτός Γενέβης. Οι δύο διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν ταυτόχρονα για να μειωθεί το κόστος και για να περιοριστεί ο προστατευτισμός. Οι δεμοί θα επιτευχθούν τελικώ τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούμε. Επίσης, πολλές από τις συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση άγνοουν το πιο σημαντικό και δυναμικό σύνορο του, του παγκόσμιου εμπορίου, του, τις νέους αναφιόμενους παίκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και οι φτωχότερες οικονομίες είναι εκείνες οι οποίες συνήθως αποκλείονται από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Τέλος, το πολυμερές εμπορικό σύστημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο λόγω της, του εύθραυστου της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχουμε δει να αναπηδούν προστατευτικές πιέσεις σε ορισμένες περιοχές. Το πολυμερές σύστημα έχει τον μοναδικό ρόλο να ανταποκρίνεται στις ε, προκλήσεις αυτές και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δύναμη. Τέλος λοιπόν, το παλί σημαίνει όχι μόνο ένα τεράστιο επίτευγμα για όλες και όλους μας, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία. Υπάρχει τώρα πραγματική πολιτική όθηση, φορά και πάνω σε αυτήν πρέπει να βασιστούμε. Μόλις τώρα άρχισε η δουλειά. Το 2014 θα πρέπει να αποδειχθεί το έτος όπου θα εφαρμόσουμε τα πρώτα αποτελέσματα μετά τις διαπραγματεύσεις και το έτος στο οποίο θα ξεκινήσει ξανά ο γύρος της Ντόχα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Όλοι έχουμε το ρόλο μας να παίξουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και αναμένω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά του ΠΟΕ. I think this Νομίζω πως το χειροκρότημα υπογραμμίζει τη σημασία της ομιλίας σας, ιδιαίτερα για το δεύτερο τμήμα, το σχεδιασμό του μέλλοντος, που ήταν ε, το, το τμήμα κλειδί της ομιλίας σας. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση, ξεκινώντας με τους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και πρώτος ο Ντανιέλ Κασπάρη από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά, που σήμερα το πρωί βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Είπατε ότι την ε, συμφωνία θέλετε να την ολοκληρώσετε μετά από ένα τάγκ ε, ε, αερίου στο Μπαλί πολλά τάγκερ με φυσικό αέριο ε, χρειάστηκαν. Ε, παρόλα αυτά καταφέρατε τη συμφωνία. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσετε να επιτύχετε και άλλα αποτελέσματα όπως αυτά που μόλις περιγράψατε. Αλλά περνώντας στην ατζέντα η μετά τον Παλί και ιδιαίτερα το θέμα της εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς διαπραγματευόμαστε με τις χώρες ΑΚΕ ε, όσον αφορά τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες. Εσείς πιστεύετε πως τώρα που υπάρχει αυτή η συμφωνία του Μπαλί, οι δικές μας διαπραγματεύσεις ε, με τις χώρες αυτές θα βοηθήσουν στην εφαρμογή των όσων αποφασίστηκαν στον Μπαλή. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή ε, μέσω της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι χώρες ΑΚΕ που κάποιες από αυτές είναι από τις φτωχότερες στον κόσμο θα μπορέσουν να ωφεληθούν στο μέλλον από το εμπόριο. Δεύτερο θέμα, είχαμε την πρώτη επέτειο της συμμετοχής της Ρωσίας στο ΠΟΕ. Και εμείς έχουμε διάφορα θέματα εδώ με τους Ρώσους, δεν είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο ε, ανταποκρίνονται στην ιδιότητα του μέλους τους στον ΠΟΕ. Διερωτώμεθα λοιπόν ποιες είναι οι δυνατότητες του ΠΟΕ από τη Γενέβη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη ώστε να στηρίξουν καλύτερα τα νέα μέλη του ΠΟΕ το καλύτερο θα ήταν νομίζω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να στηρίξουμε αυτές τις χώρες στην εφαρμογή ε, και στην ανταπόκριση μάλλον στις ανάγκες τους γιατί η ανησυχία μου είναι πως αν αρχίσουμε πάνελ και επίλυση διαφορών για όλες μας τους διαφορές με τους Ρώσους ή άλλα μέλη του ΠΟΕ δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Οπότε η ερώτηση μου είναι ποιες είναι οι στρατηγικές που έχει ο ΠΟΕ για να βοηθήσει τα νέα μέλη του ΠΟΕ να εφαρμόζουν καλύτερα τους κανόνες του. Και η τρίτη ερώτηση είναι, όταν μιλάμε για εμπόριο, συχνά μιλάμε για εμπόριο και κάτι άλλο. Ε, πώς μπορεί δηλαδή η εμπορική πολιτική να βοηθήσει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών, στην ανύψωση των κοινωνικών ε, προδιαγραφών κτλ. Και επίσης έχουμε το Σώμα Επίλυσης Διαφορών εντός του ΠΟΕ. Ε, ε, ερώτησή μου είναι... Υπάρχουν κάποιες άλλες πρωτοβουλίες με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το διεθνές, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ή άλλους για να βοηθηθούν να συστήσουν κάποιους τέτοιου μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και σε αυτούς τους θεσμούς, γιατί νομίζω όλοι συμφωνούμε ε, ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για το περιβάλλον, για τις κοινωνικές προδιαγραφές, ο ΠΟΕ μπορεί να παίξει ρόλο, ναι, αλλά δεν μπορεί να λύσει και όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι ο ΠΟΕ, τι ρόλο μπορεί να παίξει ακόμα και μετά από αυτή την επιτυχία στον Παλί, ώστε να ενισχυθούν οι πολυμερείς οργανισμοί. Έχετε υπόψη άλλες στρατηγικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, 7 πολιτικές ομάδες και ένας μακρύς ε, κατάλογος υπόλοιπων ευρωβουλευτών που θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Συντονιστής των Σοσιαλιστών τώρα, ο κύριος Μπέρντε Λάγκε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθυντά. Να έρθω σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι λίγο και αυτά που έθιξε ο κύριος Κασπάρη. Δηλαδή, εάν θεωρούμε ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά όντως αποσκοπεί στην βελτίωση των βιωτικών συνθήκων, θα πρέπει να μιλήσουμε και για κάποιες θεσμικές αλλαγές του ΠΟΕ. Για παράδειγμα και πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία. Αναφερθήκατε σε ορισμένες παραμέτρους ερωτώ μήπως χρειάζεται και κάποιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Και βέβαια και η ενδεχόμενη συνεργασία και με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας για να δημιουργηθούν κάποια πλαίσια. Και βέβαια και το ζήτημα μηχανισμών προστασίας επενδύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αυτό είναι ένα τομέα. Δηλαδή, ποιε σκέπτεστε ότι μπορεί να είναι θεσμικέ μεταρρυθμίσει. Δεύτερο, για τι διμερεί εμπορικέ συμφωνίε. Που το είπατε πολύ συμπαθητικά. Είπατε ότι υπάρχει ο ΠΟΕ, υπάρχουν και διμερεί συμφωνίε και ότι οι δυο αυτοί τομείς στην ουσία αλληλοσυμπληρώνονται. Για τη διαπραγματεύση τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών ισχύει αυτό το ίδιο ή σε ό,τι αφορά τον όγκο θα έλεγα των συναλλαγών αυτών είναι τέτοιος που θα επηρεάσει και τον ΠΟΕ. Ορισμένοι σχολιαστές λένε ότι η επιτυχία του Μπαλί κατέστη δυνατή μόνον λόγω της επικείμενης έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο εκπρόσωπος της Άλντε, ο Νικόλο Ρινάλντι. και ο Νικολό Ρινάλντι ήταν στον Παλί, όπως και ο κύριος Κασπάρη και μοιράστηκε αυτές τις ε, θαυμάσιες μέρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Γενική Διευθυντά. Εσείς καταστήσατε σαφές το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν στον Παλί και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε κρίσιμο ρόλο πριν και κατά τη διάρκεια του Παλή ώστε να είναι επιτυχής αυτή η ε, διάσκεψη. Επίσης, σύντομα αναφέρατε τη σημασία των, της κοινοβουλευτικής διάστασης ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη επικύρωση στις διάφορες χώρες. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω λίγο περισσότερο στην κοινοβουλευτική διάσταση του οργανισμού. Και αυτό είναι ακόμα ένα κρίσιμο σημείο για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα για τούτο εδώ το σώμα ώστε να γίνει απόπειρα για ανάπτυξη μιας πολύ πιο άμεσης λογοδοσίας των ε, θεσμών που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ε, συνειδητοποιώ βέβαια ότι η προτεραιότητα είναι τώρα η εφαρμογή των συμπεφωνηθέντων στο Μπαλί. Ωστόσο, Υπάρχει και ζήτημα, και το λέω αυτό ως ε, φιλελεύθερος δημοκράτης ευρωβουλευτής, Υπάρχει θέμα εξασφάλισης της καλύτερης σύνδεσης ανάμεσα στον οργανισμό του ΠΟΕ, τις διάφορες διμερείς συμφωνίες στις οποίες προβαίνουν τα κράτη-μέλη και έπειτα τους υπόλοιπους. Ποια είναι η και το κοινό. Ποια είναι η επικοινωνιακή στρατηγική που προβλέπει ο ΠΟΕ ώστε να βελτιωθεί το δημόσιο προφίλ των όσων προσπαθούμε να κάνουμε. Η κοινωνία των πολιτών κάποιες φορές είναι πολύ καχύποπτη για τι αποφάσεις, αλλά και ο επιχειρηματικό κόσμος έχει δυσκολίες από καιρού εις καιρών για να καταλάβει την καλή δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι. Και Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω στο ότι χρειάζεται να εφαρμόσουμε όχι μόνο τη στρατηγική των όσων αποφασίστηκαν στον Παλί, αλλά να εκμεταλλευτούμε και τα όσα συμφωνήθηκαν εκεί, ώστε να είναι πιο ελκυστικό το παγκόσμιο εμπόριο στις περιφέρειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο Ρόμπερ Στέρντι, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, είναι εδώ στο, στο Προεδρείο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που είστε τόσο ειλικρινείς. Έχω παρακολουθήσει τις περισσότερες ε, διασκέψεις στον Παλί και στο Χονγκ Κόνγκ και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε από τον Πίτερ Μάντελσον τι ακριβώς απέτυχε στο Χονγκ γιατί ήμασταν κοντά σε μια συμφωνία τότε και φαντάζομαι τελικά πως ήταν ε, η Γεωργία. Εσείς βλέπετε κάποια βασική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε την προσέγγιση της η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στο πακέτο του Μπαλί και προς το πακέτο του Μπαλί και τον ΠΟΕ εν γέννη. Νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο τελευταία στιγμή κινήθηκαν ε, μπροστά και η φαίνεται να είναι πιο φιλικές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αν όχι πιο φιλικές, τουλάχιστον να ενδιαφέρονται κάπως περισσότερο για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό χάρη στην Προεδρία Ομπάμα. Σε σχέση με τα όσα είπε ο Ντανιέλ, ε, συμφωνώ με τα όσα είπε, ιδιαίτερα για την κατάσταση με τη Ρωσία. Πρέπει να συνεργαστούμε και όχι να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πάνελ για ρύθμιση ε, διαφορών. Εδώ πρέπει να έχουμε μια αλλαγή στη διαχείριση, γιατί πιστεύω πως το πάνελ αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο, ε, η τελευταία λύση. Θα πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ λίγο για τη Γεωργία, γιατί Είμαστε σε έναν κόσμο όπου η γεωργία αλλάζει αυτή τη στιγμή και αυτό για να εξασφαλίσουμε αρκετές προμήθειες για να ταΐσουμε όλο τον κόσμο και με ανησυχεί που ίσως το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν που είναι γείτονες της Ινδίας μπορεί να υποφέρουν ε, ως αποτέλεσμα της ε, υποχρέωσης της Ινδίας να σταματήσει ε, την ε, πορεία της. Χρειαζόμαστε όντως μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά όχι μόνο με εσά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, αλλά και τη ΣΥΠΑ. Οτιδήποτε βοηθήσει σε, σε περισσότερη διαφάνεια μας δίνει σε όλους καλύτερη εικόνα. Ευχαριστώ. Ενωμένη Αριστερά, Ευρωπαϊκή Αριστερά, ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να πω ειλικρινά ένα θερμό καλωσόρισμα γιατί είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και η ομάδα μας ανέκαθεν τόνιζε τη σημασία του πολυμερούς συστήματος ως μια ευκαιρία και πρόκληση για όλους. Γιατί έχουμε την ε, πεποίθηση ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τα συμφέροντα των πολιτών. Πρέπει όμως να δούμε και πώς οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι είναι σε θέση να συνοδεύουν τη διαδικασία, να παρακολουθούν τη διαδικασία και εδώ, εφόσον είμαστε μαζί με την Διευθυντική Επιτροπή του ΠΟΕ, ότι η κοινοβουλευτική διάσκεψη στον Παλί ήταν κατά τη γνώμη μου σημαντική συμβολή στο να φανεί και να γίνει κατανοητό στους πολίτες ότι αναζητώνται οι λύσεις σε αυτές τις συζητήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να καταλάβουν το ΠΟΕ, να ξεπεραστεί το κενό το οποίο αυξάνεται, το χάσμα μάλλον, το οποίο αυξάνεται ανάμεσα στους φτωχού και τους πλουσίους. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις Σύμφωνα με την ε, GSE το 2030 θα έχουμε εξαντλήσει όλους τους ε, ε, πόρους μας. Ο πλανήτης μας στάνει στο, στα όρια του. Ωστόσο, ακόμα και με το πακέτο του Μπαλί, ο εστιασμός είναι στην ανάπτυξη, με ένα μοντέλο ενεργειακό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις κλιματικές αλλαγές. Ακόμα και με την ανακοίνωση ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα για τα πράσινα αγαθά, πιστεύετε ότι υπάρχει νέος προσανατολισμός για το διεθνές εμπόριο. Έπειτα, η συζήτηση ξεκίνησε στον ΠΟΕ σε σχέση με τις ισοτιμίες και το δίκαιο εμπόριο. Ε, και στην 8η διάσκεψη αντιμετωπίστηκαν, εξετάστηκαν μάλλον τα ζητήματα. Πού βρισκόμαστε, έχει υπάρξει κάποια πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενο γύρο, πρέπει να βάλω το ρολόι μπροστά, το χρονόμετρο. Κρίστοφερ Φιέλνερ, τώρα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Και επειδή πιέζει ο χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομο, Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ για την επιτυχία στο Μπαλί, κύριε Γενική Διευθυντά που είναι πολύ καλός φίλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τούμπαλιν. Οι φίλοι όμως είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Ε, Διερωτώ με λοιπόν θα μπορούσε να είναι ειλικρινής ο ΠΟΕ. Εσείς αξιολογείτε την Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική. Έχετε να υποβάλλετε συστάσεις προς εμάς, διότι εμάς μας ανησυχεί σε παγκόσμιο επίπεδο προστατευτισμός. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσέχει το ε, προστατευτισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως δηλαδή καταλήξει σε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες που θα δημιουργούσαν προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι τα πάντα. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει την εφαρμογή αυτού του πακέτου. Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. President. Welcome, General. Ο κύριος Λάχτρετ που ήταν και αυτό στον πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Ρινάλντι. Α, έφυγε ήδη. Τέλος πάντων. Της κοινοβουλευτικής διάστασης ε, το ζήτημα. Ήμουν στον πάλι στην κοινοβουλευτική διάσκεψη. Θέλω να αναφέρω το εξή. Είχα την εντύπωση ότι οι συνάδελφοι δεν ήταν τόσο ευτυχεί με τη μεταχείριση των βουλευτών στον Παλί. Δηλαδή, ούτε τι συζητήσει ε, ε, μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε ε, στην υπουργική συνάντηση, ούτε καν να τι δούμε. Και εσεί, βέβαια, σίγουρα είχατε βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά δεν μιλήσατε με του βουλευτέ. Και τελικά, ξέρετε, εμεί θα αποφασίσουμε για το πακέτο αυτό του Μπαλί. Θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ναι ή όχι. Θα πούμε ναι. ναι, εντάξει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ενδεχομένω κάποιοι θα μπορούσαν θεωρητικά να πούν και όχι. Αυτό συμβαίνει με κάποιε εμπορικέ συμφωνίε, όπω η Άκτα για παράδειγμα. πώ βλέπετε λοιπόν το μέλλον τη κοινοβουλευτική διάσταση, Δεύτερη ερώτηση, Πώ βλέπετε το ρόλο τη Ινδίας στο μέλλον, διότι είχα την εντύπωση και επειδή παρακολουθώ τα θέματα αυτά, αρχίζει να γίνεται κατάσταση όλο και πιο πολύπλοκη με την Ινδία. Δεν υπάρχει πρόθεση ή τέλο πάντων ορατή ε, πρόθεση να αλλάξει κατάσταση. Πώς ε, βλέπετε τα πράγματα. Τρίτη ερώτηση είδα ότι όλοι σας ε, οι αναπληρωτές διευθυντές είναι άρενες. Δεν θα ήταν ε, καλό να μπει και μια γυναίκα στα υψηλά αυτά κλιμάκια. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Παύλο Θάλμπα από το ΕΛΚ είναι ο ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με το Γενικό Διευθυντή ότι δεν είναι μόνος δρόμος ο ΠΟΕ για τις αγορές και ότι οι διαπραγματεύσεις και μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται και αλλού. Και δεν είναι αποκλειστική αυτή η διαδικασία του Μπάλι όμως. Αυτό που θέλω να μου πει ο Γενικός Διευθυντής είναι πώς βλέπετε ή ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπος της προόδου των συμφωνιών του Μπαλί στις διάφορες ε, διαπραγματεύσεις σημαντικών πολυμερών, περιφερειακών, ε, διμερών ε, κτλ. κτλ συμφωνιών. Ποιος είναι ο ρόλος κατά την άποψή σας των συμφωνιών αυτών στο μέλλον του Παγκόσμιου για το μέλλον θέλετε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τι μέλλον έχει το TTIP στις διαπραγματεύσεις αυτές. Επίσης, θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση που σας αφορά όχι ως Γενικό Διευθυντή, αλλά επειδή ήσασταν ε, Βραζι... Ε, βραζιλιανός, ο Βραζιλιάνος πρέσβης, ποιες είναι οι σχέσεις με το Μερκοσούρ και οι συμφωνίες του Μπαλί πώς μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις, τις πολύ σημαντικές ε, για μένα θες, σχέσεις της Μερκοσούρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, νομίζω ότι στο Βραζιλιάνο πρέσβη που είναι και εδώ ε, την συγκεκριμένα πρέσβη θα μπορούσες να θέσεις το δεύτερο αυτό σου ερώτημα, την οποία θα να καλωσορίσω κιόλα. Ε. Κάθριν Μπίρτερ από την Άλντε, επόμενη Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Ε, θα ήθελα να σας κάνω το εξής ερώτημα. Αναφέρατε είπατε ότι η Γενέβη δεν θέλετε να είναι ένα νησί αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να διαπραγματευθεί συμφωνίες εμπορικές τόσο εύκολα και γρήγορα όπως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή θα αποδυναμωθεί η θέση της Βρετανίας αν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον στον Πρωθυπουργό το νόμερο Βασίλη πρέπει να κάνει την ερώτηση σας, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος, David Campbell, ECR. Κύριε Γενική Διευθυντά, πρόσφατα ο Ρώσος πρέσβης ήταν εδώ και μας είπε πώς δραστηριοποιείται σε όλες τις επιτροπές του ΠΟΕ. Η Ρωσία. Καλή είδηση αυτή, βέβαια. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτές οι επιτροπές έχουν κάποιο ρόλο στην θέσπιση των διεθνών κανόνων και πώς μπορεί να βοηθήσει και η συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο των επιτροπών. Πρόεδρος. Ο κύριος Λάουλου από τον Μπενίν έχει το λόγο, από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω και τον Γενικό Διευθυντή του που νομίζω ότι αυτή η συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα πλούσια και γιατί πήραμε πληροφορίες σημαντικές και κυρίως γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να σας συναντήσουμε και να ε, διαπιστώσουμε το επίπεδο ε, της ε, αποφασιστικότητας, της δέσμευσής σας. Και με αυτά τα δύο στοιχεία που εντοπίζω βλέπω ότι θα πάμε πολύ μακριά μαζί. Είπατε κάποια μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, ε, τα οποία αποφασίστηκαν στον Παλί και συμφωνώ απόλυτα. Πέραν αυτών όμως χθες και μεταξύ άλλων συζητήσεων, συζητήσαμε και το σύστημα επίλυσης διαφορών σε επίπεδο ΠΟΕ σημαντικά πράγματα πρέπει να γίνουν, τα νέα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν, ο κανονισμός, μάλλον ε, η διευθέτηση των ε, διαφορών, η επίλυση των διαφορών και βέβαια και σε επίπεδο χωρών πρέπει να γίνει δουλειά, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι ε, οι χώρες είναι αυτές που θα σας εκπροσωπήσουν απέναντι στον πληθυσμό τους η κάθε μία και θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες των χωρών για το τι ε, γίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, αν μπορείτε, κατά την άποψή σας, ποιους μηχανισμούς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί και να παράσχουμε μία μόνιμη συνδρομή στις χώρες αυτές για να μπορέσουμε όλοι μαζί να εργαστούμε από κοινού. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ώρα των ερωτήσεων. Πολλές, πολλές είναι οι ερωτήσεις, πολλά είναι τα θέματα που πρέπει να θίξετε. Έχετε το λόγο. <laughs> well, a lot to answer. Πράγματι, πολλά ερωτήματα ε, πρέπει να απαντήσω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω λεπτομεριακά, θα πάνω στο επίπεδο λεπτομέρειας που θα έπρεπε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να μην ε, ξεχάσω κάποια και να απαντήσω και όσο δυνατόν πιο αντικειμενικά. Να ξεκινήσω ε, με τη σχέση μεταξύ της, των συμφωνών οικονομικής θερικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ, αν θα βοηθήσει ε, στην υλοποίηση των στόχων του Μπάλ κτλ. Ναι, πιστεύω ότι το πιστεύω απόλυτα γιατί ένας από τους στόχους της συμφωνίας ε, διευκόλυνση του εμπορίου που πετύχαμε στον Παλί είναι η ολοκλήρωση, η ενσωμάτωση των πιο φτωχών οικονομιών και στις εμπορικές ε, ροές. Πώς θα βοηθηθούν αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν στην αλυσίδα εφοδιάσμου σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα θέμα σημαντικό και θα βοηθήσει την ε, ενσωμάτωση. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα για τη Ρωσία, μπορώ να απαντήσω ίσως από κοινού αυτά. Πιστεύω ότι υπάρχει ε, μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ρωσίας, που βέβαια προσχώρησε λίγο πριν ε, από ένα χρόνο στον ΠΟΕ. Είναι σημαντικέ οι δεσμεύσει που ανέλαβε η Ρωσία. Αν δείτε το πρωτόκολλο ε, προσχώρηση τη Ρωσία, πάρα πολλέ ε, δεσμεύσει είχε αναλάβει, τι οποίε θα απαιτηθούν μεταρρυθμίσει. Θα απαιτηθούν δράσει εφαρμοστικέ στη Ρωσία και όπω και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ε, δεν είναι εύκολο να επισυμβούν οι αλλαγέ αυτέ. Θα απαιτηθεί προσπάθεια. Ωστόσο, σε ό,τι μπορώ να κρίνω μέχρι τώρα, και αυτό έχετε σε ένα άλλο ε, ερώτημα που αναφέρθηκε προηγουμένω. Είναι ε, προσιλωμένη η Ρωσία στι δεσμεύσει τη καταβάλει προσπάθειες. Υπάρχει, ξέρετε, και ένας χρόνος ορίμανσης ε, από τη στιγμή που προσχωρεί μια χώρα μέχρι ότου ε, εφαρμόσει τις αλλαγές. Και το να συμμετέχει, το να κάθεται σε μια αίθουσα, να συμμετέχει στις συζητήσεις, να ακούει τις συζητήσεις, αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Και το να καταλάβει την νοοτροπία και την κουλτούρα του αυτού οργανισμού απαιτεί χρόνο. Αλλά διαθέτουν πόρους και μέσα και ήταν πολύ υποστηρικτική η Ρωσία στον Παλί, όχι μόνο ως παρατηρητής, αλλά ενεργά. Προσπαθούσε να συγκλίνει και να βοηθήσει αυτούς που είχαν δυσκολίες να συγκλίνουν ήταν εκεί μέχρι τα πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, του Σαββάτου, συγγνώμη. Και είναι σίγουρα μια δύσκολη διαδικασία, μια πόδινη διαδικασία για όλες τις χώρες που προσχώρουν. Θα θυμάστε και τις πρώτες μέρες της προσχώρησης της Κίνας. Εκεί και πάλι ήταν αβέβαια τα πράγματα, πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση και εξελίχθηκε νομίζω θετικά. Είναι ένα μεγάλος υποστηρικτή του πολυμερούς εμπορικού συστήματος η Κίνα. Έχει ίσως κάποια προβλήματα, ίσως κάποιες τριβές και ε, το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε μεγάλο εμπορικό εταίρο βέβαια, αλλά βούληση υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τώρα την εμπορική πολιτική και πώς αυτό ε, ταιριάζει και εντάσσεται και με στις περιβαλλοντικές πολιτικές, στα κοινωνικά πρότυπα επαφή και συνομιλίες με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θέμα ήταν η εικόνα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία, τη διαφάνεια, να βελτιώσουμε την εικόνα και να είναι πιο κατανοητά αυτά που κάνουμε σε επίπεδο ΠΟΕ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μόλι μίλησα με τον ε, Guy Ryder, τον Γενικό Διευθυντή τη ε, Διεθνού Οργάνωσης Εργασία. Πριν από λίγε ημέρε είχαμε συναντηθεί δεν θυμάμαι πού, και του είπα ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε. Διότι είναι ενδιαφέρον ότι τις πιο πολλές φορές, ιδίως σε πολιτικούς κύκλους, όχι σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στο πολιτικό επίπεδο το εμπόριο θεωρείται απειλή για την απασχόληση. Και αυτό σαφώς και δεν αληθεύει. Ακόμη και από αμυγός οικονομική σκοπιά δεν αληθεύει αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν να αλλάξει αυτή την αντίληψη. Δεν λέω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την αντίθετη προσέγγιση, ότι δηλαδή το εμπόριο είναι πανάκια, λύνει όλα τα προβλήματα. Όχι. Αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα με αντικειμενική ματιά. Ποιε είναι οι προκλήσει. Πώ μπορεί το εμπόριο να βοηθήσει, να δημιουργήσει ευκαιρίες για απασχόληση άλλοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Οργάνωση εργασία ιδίω, είναι σημαντικοί οργανισμοί και θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να διασκεδάσουμε αυτούς τους μύθους. Δεν λέω να ε, έχουμε μια γλώσσα που να είναι πάρα πολύ θετική για το εμπόριο. Απλά λέω να διασκεδάσουμε κάποιους ε, μύθους, να διαλύσουμε κάποιους ε, μύθους ε, για το αν είναι καλή ή κακή η σχέση με εμπορίο απασχόλησης και τα λοιπά. Και εγώ πραγματικά θα αγωνιστώ γι' αυτό. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Έχει να κάνει αυτό, ξέρετε, και με τη διαφάνεια, με την ενημέρωση στο βαθμό που αρχίζουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο σε επίπεδο ΠΟΕ, ένα διάλογο που δεν περιορίζεται μόνο στους μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά που συμμετέχουν όλοι, όλοι όσοι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι και αυτό ήταν κάτι που πρώτη φορά γινόταν στον ΠΟΕ. Δηλαδή η διαδικασία διαπραγμάτευση έγινε με κάθε μεμονωμένη αντιπροσωπεία που καθόταν στο τραπέζι. Με την κάθε μία, όλες τις Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και α, λειτουργήσε. Απέδωσε, διότι στο τέλος της διαδικασίας μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι τελικά είδαν αυτούς ως μέλη και δικαιούχους της όλης διαπραγμάτευσης. Μπορεί να μην ήταν όλοι ευτυχεί, γιατί είναι και πολύ ε, μεγάλη αυτή η λέξη. Ήταν όμως ε, ε, ικανοποιημένοι. Είδαν ότι ωφελήθηκαν από αυτή τη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο. Η διαφάνεια, η συμπερίληψη, η ένταξη όλων, η ευκαιρία που είχαν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και πίστηκαν ότι αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτή την ίδια προσέγγιση θα συνεπάγεται αυτό μια τεράστια θεσμική μεταρρύθμιση του ίδιου του ΠΟΕ. Συμφωνίες, ε, πώς μπορούν να αντεχθούν άλλες συμφωνίες στον ΠΟΕ και τι άλλο μπορεί να γίνει κτλ. Κοιτάξτε, αν είναι αναπτυσσόμενες χώρες, οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες, όλοι τέλος πάντων, θεωρούν ότι η συμφωνία στον Παλί έχει αυτά αποτελέσματα και εφαρμόζεται, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η εφαρμογή των συμφωνιών του Μπάλι. Να δώσουμε τεχνική βοήθεια, δημιουργία ικανοτήτων, να βοηθήσουμε τι χώρε να εξυγχρονίσουν τι τελειωνικέ διαδικασίε κτλ. Εάν λοιπόν δώσουμε αποτελέσματα, φέρουμε αποτελέσματα, θα πιστέψει ο κόσμο ότι κι άλλο μπορούμε να πετύχουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει ε, καχυποψία έλλειψη εμπιστοσύνη εκ μέρου πολλών ανεπτυσσόμενων χωρών, ιδίω των φτωχότερων, οι οποίε δεν πιστεύουν πραγματικά ότι θα έχουν τη βοήθεια που τους έχουν υποσχεθεί. Άρα, καθήκον μας τώρα είναι να διαλύσουμε αυτή την καχυποψία, να τους πείσουμε. Και αν αρχίσει να ε, καθιδρείται αυτή η εμπιστοσύνη, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εισαχθούν στη συζήτηση και άλλα θέματα με τα οποία έχουν δυσκολήσει οι χώρες, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Πιστεύουν ότι στην άκρη, πίσω από την πόρτα κρύβεται απειλή, κρύβεται προστατευτισμός. Ότι θα εγκαταλείψουν το αναπτυξιακό θεματολόγιο. Βάζουμε αυτά τα νέα θέματα για να αντικαταστήσουμε την αναπτυξιακό θεματολογιο. Αυτό πιστεύουν. Άρα ο ρόλος της εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Κοινοβουλευτική διάσταση. Πολύ το αναφέρατε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ε, πιο θετικοί ε, όποτε έρχεται μια αντιπροσωπεία κοινοβουλευτική, εγώ προσωπικά την υποδέχομαι και όπου ταξιδεύω προσπαθώ να περάσω κάποιο χρόνο με τους βουλευτές. Σήμερα είμαι εδώ, είμαι στις Βρυξέλλες για αυτό το λόγο, για αυτή την επαφή. Αυτό δεν είναι υποπροϊόν ε, μιας ε, άλλης ε, επίσκεψης ή τέλο πάντων στο περιθώριο μιας άλλης επίσκεψης. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Έχω έρθει για να έχουμε διάλογο. Γιατί είναι σημαντικό. Συνειδητοποίησα ότι πράγματι στον Παλί δεν συναντήθηκα με βουλευτές για να σας πω ότι και με ειλικρίνεια δεν κοιμήθηκα πόσο να είχα χρόνο να συναντηθώ. Πέντε μέρες κοιμήθηκα οχτώ ώρες. Ήταν δύσκολες ε, οι στιγμές, ε, πράγματι δεν μίλησα, με κανέναν θα έλεγα, ε, όχι μόνο με εσάς δεν μίλησα, αλλά ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες και περιστάσεις στη ζωή του ΠΟΕ. Αυτό το επεισόδιο ήταν ένα ξεχωριστό επεισόδιο, ελπίζω να μην επαναληφθεί ή τέλο πάντων να επαναληφθεί ω προ την τελική έκβαση που ήταν θετική. Άκουσα κάποια σχόλια ότι στον Παλί δεν ε, συμμετείχα στη συζήτηση, στις διαπραγματεύσεις, ε, δεν συμμετείχατε μάλλον εσείς. Δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα, διότι κανείς δεν ε, συμμετείχε, γιατί αυτή η υπουργική διάσκεψη δεν ήταν μια διαπραγματευτική διάσκεψη, αλλά ήταν για να εγκρίνουν οι υπουργοί αυτά που έγιναν στη Γενέ. Βέβαια, είχαν μείνει κάποια ανοιχτά σημεία και υπήρχαν και πολλές ε, αγγίλες και παρενθέσεις ε, στην ε, Συμφωνία για τη διαπραγμάτευση, για την διευκόλυνση του εμπορίου. Δεν είχαν επιληθεί όλα στη Γενέβη. Πάντως δεν ήταν πραγματικά μια διαπραγματευτική διάσκεψη. Αν θέλετε πάντως συμμετοχή, αν θέλετε να συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις, αυτό δεν θα γίνει σε επίπεδο υπουργικής διάσκεψης αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας που προηγείται μιας υπουργικής διάσκεψης. Δηλαδή να μιλάτε εσείς στην περίπτωση με την Κομισιόν, τέλος πάντων άλλοι με τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Το θέμα είναι να ενημερώνεστε, να βλέπετε τι συμβαίνει και να συνεισφέρετε και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη διαφορά κατά την άποψή μου. Και το πώς εσείς ε, θα έχετε σχέση με τους ψηφοφόρους σας, με τις εκλογικές σας περιφέρειες. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά είναι η δική σας η δουλειά δεν μπορεί να φτάσει, δεν έχει τέτοια εμβέλεια, τέτοιο ευελικές. Εσεί πρέπει να μιλήσετε ε, και να έχετε επαφή με την κοινή γνώμη και να επηρεάσετε την κοινή γνώμη. Εμεί μπορούμε να το προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχουμε τον ίδιο αντίκτυπο με εσά. Δουλειά σα λοιπόν είναι να πάτε σε εκλογικέ σα περιφέρειε, ε, στον τύπο, στα μέσα, ε, στου ψηφοφόρου σα και να μιλήσετε για αυτή τη συμφωνία και να πείτε ότι είναι καλή. Και μετά τον Παλί, πάντοτε μπορεί να ακουστούν και κάποιες ε, επικριτικές φωνές που αλλιώς μπορεί να χάσουν βέβαια και τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να είναι επικριτικές κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κάποιοι που για άλλους λόγους ασκούν ε, κριτική. Πρέπει να το κάνουν. Καλό είναι αυτό. Ε, δεν έχουμε πρόβλημα. Το δεχόμαστε. Αυτές οι επικρίσεις όμως δεν απηχήθηκαν πουθενά στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Έλεγαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν σας αρέσει αυτό. Όχι, μας αρέσει απαντούσαν όμως. Το θέλαμε. Μα δεν θα πρέπει να σας αρέσει. Όχι, λυπούμε, αλλά μας αρέσει, διαφωνούμε. Μας αρέσει. Και αυτές οι επικριτικές φωνές απογοητεύτηκαν. Όμως αυτό συνέβη γιατί ήταν πάρα πολύ καλή η όλη διαδικασία, με τη συμμετοχή όλων. Έτσι, οι επικρίσεις δεν ε, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα εάν έχει γίνει σωστά η διαδικασία και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και στο μέλλον την ίδια προσέγγιση. Για τη γεωργία, για την ε, επίλυση των διαφορών, για την επιστηστική ασφάλεια, ε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, εξασφαλίζουμε την διάθεση τροφίμων σε προσιτές τιμές. Αυτά ήταν διάφορα ερωτήματα που ετέθησαν, όπως και πώς μπορούμε να παρέχουμε επαναλαμβάνω, τρόφιμα σε λογικές προσθέσεις τιμές κτλ. Ακούστε, αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε εύκολα. Είναι μια σοβαρή συζήτηση που θα χρειαστεί έναν μακρόχρονικό ορίζοντα. Δεν ε, το αντιμετωπίσαμε με δομημένο τρόπο στις διαπραγματεύσεις. Βέβαια έρχονται όλες αυτές οι πτυχές στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είχαμε μια ε, παγκόσμια και σφαιρική συζήτηση και διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα. Γιατί αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ε, επιστημιστική ασφάλεια κλείνοντα κάποιε αγορέ, μπορεί να δημιουργήσουμε κάποια προβλήματα, να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε άλλε χώρε. Η επιστημιστική ασφάλεια του ενό ε, συχνά δημιουργεί επιστημιστική ανασφάλεια σε κάποιον άλλο. Άρα αυτή η ισορροπία που πρέπει να βρεθεί είναι λεπτή και τα συζητήσαμε. Στον Παλ... Η Ινδία είχε μια πρόταση, δηλαδή, ε, μάλλον και τη στήριξαν και άλλε αντισόμενες χώρε, αλλά πολλέ αντισόμενες δεν τη στήριξαν. Γιατί ακριβώ υπάρχει αυτό το θέμα τη ισορροπία. Μια επιστημική ασφάλεια σε μια χώρα μπορεί να είναι επιστημική ανασφάλεια σε μια άλλη. Άρα πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική συζήτηση που δεν έγινε σε επίπεδο ΠΟΕ. Υπάρχουν και άλλα βήματα συζήτηση, ΦΑΟ, κτλ. Συμφωνώ με όσους όμως θεωρούν ότι θα πρέπει να βαθύνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Για άλλες πρωτοβουλίες, ε, πρέπει να συζητήσουμε Greenwoods, περιβάλλον, πράσινα δάση, εμπορικά συμφέροντα εταιριών ή τομέα της οικονομίας. Δεν είναι μη συγκοινωνούνται αυτά τα δοχεία κατά ανάγκη, μπορεί και να συγκοινωνούν. Και υπάρχει αυτή η καχυποψία που είπα και πριν. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια πιο εμβαθυμένη, μια πιο εισβάθος συζήτηση. Τώρα, συστάσεις για την ευρωπαϊκή Μπορική πολιτική, φυσικά και δεν έχω καμία σύσταση να διατυπώσω, πέραν από μια παράκληση στηρίξτε ε, το πολυμερές εμπορικό σύστημα του ΠΟΕ. Θα το κάνουμε λοιπόν πρώτα. Ωραία, πολύ ευχάριστο αυτό. Για να δω τι άλλο για την Ινδία. Η Ινδία νομίζω ότι είναι σε μια ε, κάπως ιδιόμορφη κατάσταση, τεράστιος ο πληθυσμός, μεγάλο ποσοστό πολύ φτωχοί άνθρωποι, προβλήματα με την ε, ασφάλεια των τροφίμων, προσπαθούν και αυτοί όπως και άλλες ανεψόμενες χώρες να αναπτυχθούν. Νομίζω ότι η συμμετοχή της Ινδίας στο πολυμερές εμπορικό σύστημα είναι όσο σημαντική όσο και η συμμετοχή οποιασδήποτε άλλη αναπτυσσόμενη χώρα των ίδιων διαστάσεων, του ίδιου μεγέθου. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και τι δυσκολίε και τι ευαισθησίε, αλλά και τι ευκαιρίε που θα έχει και η ίδια η χώρα αν συμμετέχει στι πολυμερεί διαπραγματεύσει. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα εάν ακούμε ένα τον άλλο. Στον Παλί έτσι έγινε. Και είδατε το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, μεροληψία ως προς το φύλλο ε, των συνεργατών μου, ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξω τους συνεργάτες μου γιατί ήταν όλοι με πολύ ψηλά προσόντα. Εσείς που είστε πολιτικοί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί κανείς να κάνει. Όταν προσπαθεί να εξεύρει ισορροπία μεταξύ ε, των προσόντων, των ικανοτήτων και υπήρχαν πολλές γυναίκες υποψήφοι που θα μπορούσαμε να είχαμε ε, συμπεριλάβει. Αλλά δεν το, επέλεγε, δεν το ε, επέτρεψε η διαδικασία επιλογής και η Επιτροπή Επιλογής αν θέλετε. Αν εγώ, αν υπάρχει κάποιος που θεωρώ ότι μια γυναίκα μπορεί να αναλάβει τα ενία του κόσμου, είμαι εγώ. Γιατί η γυναίκα μου, οι κόρες μου, είναι και οι δύο γυναίκες. Και έχω και δύο εγγόνες. Άρα είμαι μεγάλος ένθερμος ε, υποστηρικτής της γυναικής παρουσίας ε, στους κύκλους ε, λήψης αποφάσεων. Και στο δικό μου γραφείο, από τις έξι συνεργάτες μου, οι τέσσερις είναι, είναι γυναίκες. Αν είσαι και γυναίκα μου, αλλά τέλο πάντων κατάλαβε ότι είναι βοηθή μου γιατί είναι πάρα πολύ καλές στη δουλειά τους. Ε, υπάρχει λοιπόν τουλάχιστον εκ κάποια μεροληψία. Τώρα, για το TTIP και άλλες μέρες συμφωνίες ε, μίλησαν συντομία. Συμπληρωματικά με αυτά που κάνουμε στον ΠΟΕ, είναι, αυτά, είναι αυτές μάλλον συμφωνίες. Το θέμα είναι να μην εστιάζουμε εκεί και να ξεχνάμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Γιατί αν δεν προχωρήσει και το πολυμερές, τελικά θα πολλαπλασιαστούν τα πρότυπα και οι κανόνες μέσω αυτών των διμερών συμφωνιών. Και θα υπάρχουν πολύ περισσότερες απαιτήσει για την εμπορία των προϊόντων. Τελικά λοιπόν... Θα είναι σαν να έχουμε ε, ένα μπολ με μακαρόνια, όπως το είπαν κάποιοι, ε, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλούς κανόνες ε, κατακαιρματισμένους, ε, διαφοροποιημένους. Όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να βαδίζουμε παράλληλα, γιατί αν όχι θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα ότι είναι πολύ μεγάλη η πρωτοβουλία και πώς αυτό θα επηρεάσει τους πολυμερείς κανόνες. Κοιτάξτε, στο βαθμό που οι τεράστιες αυτές οι οικονομίες μπορούν να συμφωνούν σε κάποιους τομείς, αυτό μπορεί να βοηθήσει και το πολυμερές επίπεδο, γιατί πολλά διέξοδα που έχουμε στο πολυμερές σύστημα περιέχονται από τους μεγάλους πρωταγωνιστές που δεν έχουν σύμφωνη γνώμη σε τεχνικά πρότυπα, ε, υγειονομικά, φυτογειονομικά, τρίψ, ε, τεχνικούς φραγμούς κτλ δασμούς δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να βοηθήσουν οι συνομιλίες και στο πολυμερές σύστημα. Γιατί λοιπόν να μην το δούμε και θετικά. Αυτό που ελπίζουμε να μην συμβεί είναι να δημιουργηθούν οχυρά. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο όμως, ιδίως ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές, γιατί μιλάμε για οικονομίες που έχουν ήδη πολύ χαμηλούς δασμούς γενικά, όχι παντού, γενικά. Για να δω τι άλλο. Σίγουρα θα μου διαφύγουν κάποια ερωτήματα, κάνω ό,τι μπορώ για να καλύψω τα πάντα. Ε, και αυτό που είπα ε, έχουν να κάνουν με την ε, συμμαχία του ειρηνικού, τις χώρες ΑΚΕ και όλους. Πρέπει να είναι υποστεκτική ως προς τον ΠΟΕ και το πολυμέρες εμπορικό σύστημα, όλοι αυτοί. Πιστεύω ότι περισσότεροι θα είναι. Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, αν θα συμμετέχει ανεξάρτητα ή σε μια ομάδα. Αυτή είναι απόφαση του Ηνωμένου Βασίλειου. Δεν μπορώ να την πάρω εγώ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, όσο περισσότερο ένα κράτος ε, μπορεί να στηρίξει ε, και να επερασπιστεί ένα θεματολόγιο, ε, μια υπόθεση, ένα στόχο μέσα σε μια ομάδα, τόσο πιο μεγάλη μεγάλης πάντως έχει. Αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να σας πω, να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Γιατί η Ρωσία την ανέφερα ήδη, προσπάθησα να απαντήσω. για την επίλυση διαφορών, για τις πιο φτωχές χώρες και πώς μπορούν να ωφεληθούν, πώς μπορούν να συμμετέχουν. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μια μεγάλη πρόκληση διότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών δεν σχεδιάστηκε για, τακτικά, για τα τακτικά μέλη του ΠΟΕ αλλά για να βρεθεί μια διέξοδος σε, στο πρόβλημα που υπήρχε μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών που ήταν διαιρεμένοι και διχασμένοι. Αν οι συστάσεις επιτροπής δεν εφαρμοστούν, στο τέλο τη δικασία τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις, να εξουσιοδοτηθεί, μάλλον να εγκριθούν κυρώσεις προ ένα μέλος. Αλλά αν έχουν μια τεράστια οικονομία, ε, και αν υπάρχει ασυμμετρία, δηλαδή αν κερδίζει μια πολύ φτωχή μικρή χώρα την ε, διαφορά απέναντι σε μια τεράστια υπερδύναμη, ουσιαστικά αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, διότι ε, θα επιβάλλει αντίπεινα η μεγάλη χώρα. Άρα είναι σαν να πυροβολεί η μικρή χώρα το ίδιο της το πόδι. Με όλες τις ατελείες του όμως το σύστημα μέχρι τώρα λειτουργεί. Λειτουργεί σχετικά καλά. Περισσότερο από το 90% των πορισμάτων και των συστάσεων έχουν εφαρμοστεί. Ένα 10% δεν έχει. Τα κράτη-μέλη όμω είναι σε διαπραγματεύσει, συνομιλούν μεταξύ του για να βρουν μια λύση. Στι περισσότερε περιπτώσει όμω έχει λειτουργήσει καλά το σύστημα. Προσπαθούμε οι λιγότερο ανεπτυγμένε και οι αναπτυσσόμενε χώρε να συμμετέχουν περισσότερο, να εξοικειωθούν περισσότερο με το σύστημα, να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν. Κάποιε χώρε το έχουν χρησιμοποιήσει και επειδή μιλώ για ασυμμετρίες, είχαμε μια υπόθεση αντίγουα μπαρμπούντα ε, κατά ΙΠΑ. Καταλαβαίνετε βέβαια πόσο δύσκολη ε, ήταν ε, αυτή η κατάσταση λόγω της ασυμμετρίας σε ό,τι την οικονομική δύναμη. Πάντω μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να συμμετέχουν περισσότερο αυτέ οι χώρε. Μία από τι δυσκολίε είναι, για παράδειγμα, η οικονομική πόρη. Διότι οι υποθέσει αυτέ δεν είναι και ολιγοδάπανε είναι πάρα πολύ δαπανηρές και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε τρόπους να δοθεί βοήθεια, να δοθεί εκπαίδευση που ε, χρειάζονται οι χώρες αυτές. Διότι δεν έχει νόημα οι χώρες αυτές να αναπτύξουν έναν όλο στρατό από δικηγόρους ε, κτλ. Γιατί μπορεί μία φορά στα 15 χρόνια να χρειαστεί να καταφύγουν σε αυτό το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την κατάσταση και να είμαστε δημιουργικοί. Δεν είναι εύκολο και ίσως αυτό είναι ένα από τα ελαττώματα μέσα στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Δεν υπάρχει πραγματική συμμετρία, δεν μπορούν να, να συμμετέχουν ισότιμα και εξίσου αποτελεσματικά οι μικρές και οι μεγάλε χώρε. Δεν απαντήσατε για τη σημασία των επιτροπών, κύριε, και τη Ρωσία και τη συμμετοχή της Ρωσίας στις επιτροπές, ε, πόσο σημαντικό είναι να είναι δραστηριοποιημένη η Ρωσία Απάντηση. Ναι, συμμετέχει η Ρωσία σε επιτροπές πράγματι και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό οι χώρες να αντιλαμβάνονται τις δεσμεύσεις τους. Εκεί γίνεται και η αξιόλες από ομοτήμους, όπως το λέμε, εκεί γίνεται η διάδραση, η αλληλεπίδραση και ρωτάμε τι χώρε, για πείτε μα πώ αυτό συνάδει με τι δεσμεύσει, σα και τι περισσότερε φορέ ο πρέσβη ή ο εκπρόσωπο πρέπει να πάει στην πρωτεύουσά του και να πει κοιτάξτε, κάνετε το τάδε, το δίνα, αλλά εδώ εμένα με ρωτάνε αν αυτό συνάδει με τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει. Πώ θα του εξηγήσουμε αυτά που κάνουμε. Και τι περισσότερε φορέ, αυτό βοηθά και τι ίδιε πρωτεύουσε να κατανοήσουν ότι τις παρακολουθούν, τις ελέγχουν οι υπόλοιποι και ότι τελικά εάν δεν προσπαθήσουν ε, να υλοποιήσουν τα συμπεφωνημένα μπορεί να είναι ε, αντικείμενο μονομερών κυρώσεων ή αντικείμενο μιας διαφοράς να μπουν στο μηχανισμό επίλυσης διαφόρων κτλ. Δεν θα έβαζα ένα ποσοστό, αλλά θα, ας πω ένα 90% τουλάχιστον. Πιστεύω των τριβών και των ε, ανησυχιών και των προβλημάτων να αντιμετωπίσουν στο επίπεδο των επιτροπών. Η επίλυση διαφορών είναι το ε, τέλος, το τελευταίο στάδιο, αφού ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία των επιτροπών κτλ. Τότε φτάνει, Τότε φτάνει κανείς στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Αυτό είναι σημαντικό να συμμετέχει ανεργά σε επιτροπές η Ρωσία. Αυτό είναι σημαντικό πράγματι. Ρομπέρτο, μπορείς να συνεχίσεις με βάση τα όσα είπε ο Ρόμπερτ Στέρντι για τη θέση των ΙΠΑ σε σχέση με την ΤΟΧΑ. Τι, εμείς πιστεύαμε πως η Ντόχα είχε πια πεθάνει η διαδικασία της Ντόχα. Ε, ενώ η φαίνεται φαίνεται να είναι πιο θετικές αυτή τη στιγμή για να αναζωογονηθεί η Τόχα. Ποια ήταν η αντίδρασή τους. Γιατί νομίζω πως είναι θέμα κλειδί. Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς τη ΣΥΠΑ τώρα, ό,τι και να λέμε. Μπορείς, είσαι βέβαιος ότι ε, έχουν κάποια νέα στάση ή είπα σε σχέση με αυτό. Να, συγγνώμη, ναι, ξέχασα αυτή την ερώτηση γιατί ε, στον κατάλογό μου δεν την είδα καλά. Ε, κοιτάξτε, οι Αμερικανοί στο Μπαλί έδειξαν πολύ μεγάλο βαθμό δέσμευση ήθελαν να προχωρήσουμε και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τα καταφέρουμε. Ο Μάικλ Φρόμαν ήταν πολύ δραστήριος. Πέρασα περισσότερες βραδιές μαζί του στον Παλί παρά με τη σύζυγό μου. Δεν είναι και πολύ καλός ιονός αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την επίτευξη της επιτυχίας. Ε, Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό η αμερικανική, ο βαθμός μάλλον ε, της αμερικανικής δέσμευσης ε, εξαρτάται από το γεγονός ότι πίστευαν πως μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Αυτό πίστευαν. Πίστευαν πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ιδιαίτερα μετά το 2008 Είδα μια αποστασιοποίηση από τις διαπραγματεύσεις της Γενέβης από πλευράς των Αμερικανών. Εγώ πιστεύω και εδώ σας δίνω την προσωπική μου άποψη πως σε μεγάλο βαθμό λόγω της δυσπιστία τους γιατί πίστευαν δηλαδή ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Εφόσον δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα, γιατί να ασχολούμεθα να, να σπαταλάμε χρόνο για κάτι που δεν πιστεύουμε ότι θα επιτύχει. Και γι' αυτό και άρχισαν να διερευνούν τις πολυμερείς, άλλου είδους συμφωνίες, αλλά κυρίως όπως σας είπα, λόγω του ότι ε, δεν πίστευαν ότι ήταν βιώσιμη η πολυμερής ε, συμφωνία. Νομίζω πως όλα αυτά έχουν αλλάξει. Εγώ συνομιλώ μαζί τους ε, διαρκώς από τον Παλί ήταν πολύ θετική ε, μέχρι στιγμής. Και όλες αυτές οι παράμετροι που σας ανέφερα τις δέχονται. Δέχονται και λένε ότι είναι πρόθυμοι να δεργαστούν από αυτές τις βάσεις. Είπαν ότι ναι, θα, είμαστε, θα έχουμε ανοιχτό μυαλό, θα διερευνήσουμε τις ιδέες, δεν είμαστε προσκολλημένοι σε οτιδήποτε. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Το, μόνο μήνυμα δηλαδή που κατάλαβα εγώ ήταν να μην ξαναπέσουμε στις κακές συνήθειες. Και ποιες είναι οι κακές συνήθειες για αυτούς? Η αποτυχία. Να μην ξαναβρεθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου διαπραγματευόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα διέξοδο, αλλά να το ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Στο βαθμό που μπορούμε να δείξουμε, όχι μόνο στους Αμερικανούς, αλλά σε όλους, ότι έχουμε ένα στόχο επί, ε, απτό ε, ότι είναι σοβαρό και ότι όλοι συμφωνούν να το κάνουμε αυτό και πριν τον πάλι ήταν ε, ασαφές ότι όλοι θέλαμε να γίνει αυτό πιστεύω πως θα έχουμε επιτυχίες και ότι θα μπορέσουμε να δούμε και ευελιξία και δέσμευση που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέχρι ε, τέλος, σε έκβαση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέω Πριν να σας αφήσω να φύγετε, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις. Φυσικά ήταν εξαιρετική εκδήλωση σήμερα. Είμαστε, είναι μεγάλη μας τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ και πιστεύω ότι ανταποκριθήκατε στις προσδοκίες μας απολύτως. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ε, στηρίξω όταν λέτε ότι προσεκληθήκατε από το κοινοβούλιο μας και γι' αυτό βρίσκεστε εδώ. Να σας πω ότι συναντηθήκαμε πριν από κάποιες εβδομάδες και θα θυμίσω, θύμισα μάλλον στον ε, Ρομπέρτο, ότι ήταν εδώ στις Βρυξέλλες, όταν είναι υποψήφιος για τη θέση την οποία τώρα κατέχει, εγώ του είχα πει ότι εάν τελικά εκλεγείς, πράγμα που ελπίζω να γίνει, θέλω την δέσμευσή σου ότι θα έρθει στην Επιτροπή μας, όσο γίνεται πιο σύντομα. Έχουμε προσωπικά συναντηθεί πριν από κάποιες εβδομάδες και του θύμισα αυτή τη δέσμευση και του είπα, στην ουσία τον υποχρέωσα να ανταποκριθεί στην ε, υποσχεσή του, αλλά ανταποκρίθηκε, όπως είπα, με αφελή τρόπο. Δεν χρειάζεται να με αναγκάσεις. εγώ συνήθω τηρώ τι υποχρεώσει μου και τι δεσμεύσει μου. Ωραία λοιπόν το είπα τότε, α βρούμε μια ημερομηνία. Και ειλικρινά πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ καλή ε, αρχή για τι σχέσει ανάμεσα στη νέα Γενική Διεύθυνση του ΠΟΕ με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μα τώρα και στο μέλλον. Διότι είμαι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για μια ε, και μοναδική φορά που έρχεσαι. Ε, εδώ είπαμε ότι ως ήθιστε η επόμενη μας συνάντηση θα είναι στη Γενέβη με την ευκαιρία του Public Forum, του Δημοσίου φόρουμ του ΠΟΕ και θα συμμετέχουμε εκεί δραστήρια όπως συνηθίστε γιατί είναι ένα από τα πιο ωραία, τις πιο ωραίες εκδηλώσεις για να φτάσουμε στους, στο κοινό, στις ΜΚΟ και στους διάφορους φορείς και είμαστε δραστήριοι ε, δραστήρια μέλη. Δεν θέλω να το ξαναπώ γιατί πιστεύω πως τα πράγματα είναι αρκετά ε, σίγουρα ότι το δικαίωμα το οποίο μας είχε δοθεί στον προκάτοχό σας να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε τους χώρους του ΠΟΕ, θα το έχουμε και πάλι. Και ότι θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε και να παρακολουθούμε τη steering committee. Το των Λευθέντων ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τα όσα είναι κοινά, αλλά και για να μάθουμε ποιες είναι οι προσδοκίες, οι ελπίδες και τα σχέδια για το μέλλον για τον ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.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 Colleagues, the ναι, Τελείωσε το διάλειμμα αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα τώρα της ημερησίας διατάξεως σύντομη παρουσίαση της εκθέσεως της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην ε, Διευπουργική Διάσκεψη του Μπαλί. Την έκθεση την έχετε στους φακέλους σας. Η αντιπροσωπεία μας είχε διτό στόχο και να παρακολουθήσει την ε, Διευπουργική Διάσκεψη κάτι που αποδείχθηκε απολύτως συναρπαστικό διότι παρακολουθήσαμε προσεκτικά τις, τις διαπραγματεύσεις και εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μάλλον τα όργανα αυτά μας τήρησαν πλήρως ενημέρους για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για άνευ προηγουμένου περίπτωση όπου συμμετείχε και το Κοινοβούλιο εκτός από τις εκπροσώπες της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Πρόκειται για αλλαγή της τάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και βεβαίως καλοδεχούμενη. Έχουμε συνηθίσει να επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν αυτό βεβαίω είναι όρθο, αλλά θα πρέπει επίσης ορθό να είναι να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καλώς έπραξε. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν να συμμετάσχουμε στην ε, συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΠΟΕ. Ο Ρομπέρτο Βέντο δεν μπόρεσε να έρθει στην συνάντησή μας. Έστειλε ωστόσο έναν από τους αναπληρωτέ γενικούς διευθυντές, ο οποίος ε, ήρθε δύο φορές και έτσι και από την άποψη αυτή λοιπόν δεν μπορούμε να παραπονηθούμε σε ό,τι αφορά την στάση της ηγεσίας του ΠΟΕ. Έχετε την έκθεση, στα αγγλικά έχει δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα και έχετε τη δυνατότητα τώρα να ε, κάνετε σχόλια, ή παρατηρήσεις έχετε, παρατηρήσεις. Ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ. Δύο σύντομα σχόλια. Κάτι που με εξέπληξε ήταν πως συνεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Δεν είμαι από εκείνους που είμαι συνήθως ευγενής ιδιαίτερος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην περίπτωση αυτή πραγματικά ε, αποδείχθηκαν πολύ συνεργάσιμοι. Το δεύτερο είναι τα όσα θα εφαρμόσουμε στο μέλλον, και αυτά συζητήσαμε βέβαια και με τον Γενικό Διευθυντή πριν από λίγο, είναι αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση και η σημασία της σε όλες τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα. Εμείς αποδείχτηκε ότι ήμασταν προνομιούχοι απέναντι στους εθνικούς βουλευτές και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε ώστε να ενισχύσουν και αυτοί το ρόλο τους. Το δεύτερο και το τρίτο σχόλιο τώρα είναι ότι θα ήθελα να πω ότι μας υποστήριξε θαυμάσια το προσωπικό που ήταν παρόν. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους όσοι συνεργάστηκαν ε, μαζί μας στην περίπτωση εκείνη. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Βιτάλ Μορέιρα. Ευχαριστώ που θυμήσατε και το πραγματικά αξιόλογο έργο του προσωπικού. Όλες και όλοι ανεξαιρέτως συνεργάστηκαν θαύμασια. Άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ λοιπόν. Συμφωνώ μαζί σας, Γιώργ. Και μακάρι και όλοι οι εθνικοί βουλευτές που ήταν στον Παλί να είχαν τη δυνατότητα της ίδιας εμπλοκής με τον που ε, μας ζήλεψαν βεβαίω για τη δική μας ικανότητα να ενσωματωθούμε και βεβαίως να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, το οποίο υπό Λιθουανική Προεδρία ήταν πραγματικά, ε, αποδείχθηκε εξαιρετικά θετικό. Ωραία. Το επόμενο είναι το θέμα 6, όπου προβλέπεται συζήτηση με συμμετοχή των δύο μιζώνων ενδιαφερομένων, κοινωνικών εταίρων δηλαδή, business community και ευρωπαϊκών εργατικών συνδικάτων. Καλωσορίζω την κυρία Μπερναντέτ Σεγκό, Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων και επίσης την κυρία Ντοσάντος ε, από την οργάνωση Business Europe Πρόκειται για μέρος της τακτικής αυτής επαφής μαζί των και τώρα που προσεγγίζουμε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας είναι χρήσιμο να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με στόχο να συζητήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες, να ακούσουμε ποια είναι η αξιολόγηση στην οποία προβαίνουν οι οργανώσεις τους για το στάδιο που βρισκόμαστε και για το πώς θα προχωρήσουμε. Η κυρία Σεγκό πρώτη. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Μα σας έψαχνα αλλού. Καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ε, και κάποια ευκαμψία μπορώ να δείξω βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Γαλλικά για να ακουστεί και κάτι άλλο. Με μικρόφωνο όμως. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων, την οποία προσωπώ εδώ, για να σας μιλήσει. Η Συνομοσπονδία μας αντιπροσωπεύει τα εργατικά συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ε, πιο ευρέως στην Ευρώπη αλλά και τις κλαδικές οργανώσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς δραστηριότητας. Είναι σαφές ότι για μας η εμπορική πολιτική έχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ότι αυτό το ενδιαφέρον αναπτύχθηκε κυρίως από την δημιουργία του Global Europe, της πολιτικής για μια παγκόσμια Ευρώπη το 2006, όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιταχύνει την δέσμευσή της σε εμπορικές συμφωνίες διμερούς ή διπεριφερειακού τύπου. Το ενδιαφέρον μας αυξήθηκε μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας που αύξησε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως για τα θέματα επενδύσεων και που έδωσε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Ε, παραδοσιακά στηρίξαμε την προσέγγιση, ή μάλλον τις πολυμερείς προσεγγίσεις ε, στις εμπορικές πολιτικές, ωστόσο έχει καταστεί αρκετά σαφές και παρά τις προσπάθειες του κυρίου Αζεβέντο που μόλις ε, σας απευθύνει το λόγο και τις προσπάθειες του Πασκαλαμή πριν, ε, του προκατόχου του, κατέστη σαφές για μας ότι ο κόσμος του εμπορίου έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο υπερβολικά περίπλοκος για τον ΠΟΕ που δεν κατάφερνε πραγματικά να επιτύχει τους στόχους του και δεν είχε και τα μέσα στη, που χρειαζόταν στη διαθεσή του. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι παρά τις προσπάθειές μας, παρά τις προσπάθειες των συνανθέλφων του Διεθνούς Συνδικαλιστικού Κινήματος που στόχο έχουν να δοθεί μια κοινωνική διάσταση στις εμπορικές συμφωνίες και επιμένουμε ώστε αυτή η διάσταση να υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ωστόσο πως υπάρχει μεγάλη αντίσταση από πλευράς ε, πολλών χωρών του ΠΟΕ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πέρα από κάποιες κοινέ μελέτες με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. άκουσα τον κύριο Ζεβέντο που είπε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Γκάι Ράιντερ. Ελπίζω πως θα έχει κάποια περισσότερα μάλλον πιο από τα αποτελέσματα από ό,τι μέχρι σήμερα. Παρακολουθήσαμε τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες ε, του κοινο... Ε, ε, εμπορικές θα πρέπει να και μάλλον θα πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα σε εμπορική συμφωνία και συμφωνία σύνδεσης. Ξέρω ωστόσο ότι η δύναμη μόχλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο ισχυρή στον εμπορικό τομέα από ότι σε άλλους τομείς όπω α πούμε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης παρά τις προσπάθειες ε, αυτής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, τις οποίες χαιρετίζω, είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα της δράσης στον τομέα του εμπορίου είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε πολλούς άλλους τομείς. Το άρθρο 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρίζει ότι η δράση, και το έχω στα αγγλικά, αλλά λέει ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή ε, θα πρέπει να καθοδηγείται από, αρχές, από τις αρχές που ενέπνευσαν την ίδια της τη δημιουργία και την ανάπτυξη αλλά και τη διεύρυνσή της. Ε, είμαι βεβαία πως δεν χρειάζεται να παραθέσω ολόκληρο το άρθρο Πάντως η ιδέα είναι ότι η εμπορική πολιτική καλύπτεται από αυτές τις προθέσεις και θα έπρεπε να καλύπτει τα ιδεώδη τα οποία που ε, αντιπροσωπεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εμπόριο μπορεί να δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Δεν λέω το εμπόριο δημιουργεί, λέω ότι δύναται να δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Μπορεί να δημιουργήσει θέσει απασχόληση, Άκουσα και τα όσα είπε ο κύριο Ζεβέντο σε αυτό το, για αυτό το θέμα. Ε, δυνητικά λοιπόν είναι αληθές, αλλά δεν αληθεύει πάντα. Η... τα ευρωπαϊκά κράτη είναι εμπορικά κράτη και δεν έχω καμιά αμφιβολία πως η Ευρώπη μπορεί να είναι καλός ανταγωνιστής σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο εάν υπάρχει ε, ισορροπημένο εμπόριο. Ως ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων είμαστε αντίθετοι με τα προστατευτικά αισθήματα που προωθούνται από ακραίες πολιτικές ε, και από τα πολιτικά άκρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής ε, περίοδου. Τα αισθήματα αυτά είναι αντιπαραγωγικά από οικονομικής άποψης και φλερτάρουν με την ξενοφοβία. Όμως ε, απορρίπτουμε επίσης την ιδεολογία του ελεύθερου εμπορίου που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ε, κοινωνικές συλλογικές μας προτιμήσεις ε, που συνοψίζονται μέσα στην ιδέα και την έννοια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Και εδώ χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα για την εισαγωγή αναφορών για την παρατήρηση των περιβαλλοντικών και εργατικών προτύπων διεθνούς επίπεδου για τις περιπτώσεις ε, του κοινωνικού ντάμπινγκ, καθώς και για τη δυνατότητα που δίνεται στα συνδικάτα και άλλα ως εμπλεκόμενος να υποβάλουν καταγγελίες, να καταθέτουν καταγγελίες. Και ευχαριστώ και όλους όσους εδώ στο Κοινοβούλιο στήριξαν αυτές τις τροπολογίες. Ελπίζω πραγματικά πως ε, οι τροπολογίες αυτές θα οδηγήσουν προς ένα θετικό τριμερή διάλογο γιατί δεν θα αντιστραφούν. Το εμπόριο θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς απασχόλησης. Αυτός είναι ένας στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αν ξεχαστεί θα έβαζε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο κίνδυνο, διότι οι πολίτες που θα ψηφίσουν δεν θα το ξεχάσουν αυτό και αυτό με οδηγεί να μιλήσω για το dip μιλώ για το σύντμηση στα αγγλικά και γύρω από αυτό το θέμα αποκρισταλώθηκαν οι οι συζητήσεις, αν και δεν είναι η μοναδική συμφωνία που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε πεπισμένοι από τα νούμερα τα οποία διανεμήθηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη και τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι προτάσεις, μάλλον οι, η πρόταση που λέει ότι αυτή η ίδια συμφωνία μόνη της μπορεί να μας βγάλει από την κρίση δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θέλουμε ένα νέο σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη και αυτό πρέπει να γίνει με βάση τις γραμμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων. Χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική η οποία να ενσωματώνει τις τους προβληματισμούς του διεθνούς εμπορίου. Και αναγνωρίζω κύριε Πρόεδρε πως είναι ίσως μια ανάλυση συζήτηση αυτή που ελπίζω όμως ότι θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Εν πάση περιπτώσει, αξιολόγηση του αντικτύπου νομίζω πως είναι απαραίτητη οπωσδήποτε, διότι θα πρέπει να μας πούν ποιες θέσεις απασχόλησης θα μπορέσουν να δημιουργηθούν, με τι μισθούς και σε ποιες συνθήκες θα πρέπει να μας, πείτε σε ποιους, να μας πούνε μάλλον σε ποιους τομείς και σε ποιες περιφέρειες θα δημιουργηθούν αυτές τις απασχόλησεις. Και είναι σαφές ότι ζητάμε και μέσα προσαρμογής. Ορισμένοι πρότειναν να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αλλά για να τα πω στα γαλλικά, να τα πω ξεκάθαρα, το Ταμείο αυτό δεν είναι στο ύψος των απαιτήσεων, των όσων δηλαδή θα χρειαστούν. Για μας οι αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης είναι ένα θέμα κλειδί, υπάρχουν και άλλα, αλλά εγώ θα θίξω μόνο ορισμένα. Ζητάμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Και γι' αυτό έχουμε και ήμασταν επικεφαλής των διεκδικήσεων. Και τώρα ακούγονται κάποια πράγματα από πολιτικής άποψης ε, σχετικά και χαιρετίζουμε την απόφαση της Κομισιόν πρόσφατα να δημοσιεύσει κάποια από τα έγγραφά της και να δημιουργήσει μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία περιλαμβάνει τα συνδικάτα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης είναι πρόοδος, αν και έγινε ε, υποποίηση για την Κομισιόν, όταν δηλαδή ανακοίνωσε ότι θα γινόταν μια διαβούλευση για την ρύθμιση διαφορών ανάμεσα στους επενδυτές και τη χώρα και τις χώρες. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με τον Επίτροπο Τεκούχτ προσφάτως, αλλά χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Ένα όχι σε αυτόν τον κανονισμό για τη ρύθμιση των διαφορών θα μεταφραστεί ως, ως όχι στις διαπραγματεύσεις ή έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα απλό κάλυμα που θα επέτρεπε στην Κομισιόν να δημοσιεύσει ή να θέσει επιχάρτου την συμφωνία για ρύθμιση διαφορών που είναι επιτόπιτος και που έχει ήδη συμφωνηθεί με τον Καναδά. Όπως και άλλοι πρόεδροι είχα τη δυνατότητα να εξετάσω τις ε, οδηγίες ε, για τις οποίες διαπραγματεύεται η Κομισιόν και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλοί, πολλές αμφιβολίες, όχι απλά δισταγμοί, αλλά αμφιβολίες των κρατών μελών για να ε, ακολουθήσουν αυτούς τους μηχανισμούς ρύθμισης διαφορών. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν να είναι βασιλικότερη του βασιλέως και να συνεχίζει να ασκεί ώστε να ε, δημιουργηθεί ένας τέτοιος ειδικό μηχανισμός και επί την άποψη της διαφάνειας. Γιατί η εντολή της Κομισιόν δεν κατέστη δημόσια δεν δημοσιεύτηκε. Από τα όσα γνωρίζω, η Γερμανία ήταν επικεφαλής αυτής της αντίθεσης ε, δημοσίευσης της εντολής και αυτό που ε, είναι παράξενο είναι ότι την πλευρά της, ε, των ΗΠΑ είδαμε αυτήν την εντολή, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια της NSA. Γιατί λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση και εφόσον δεν γίνεται να διαβουλευτεί κανείς για τους μηχανισμούς ρύθμισης των διαφορών, γιατί να μην μπορεί να διαπραγματευτεί για άλλες ε, πτυχές οι οποίες είναι εξίσου ευαίσθητες. Ναι, μάλιστα, μάλιστα, συντομεύω. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα και που αγγίζει άμεσα την απασχόληση και θέλουμε να είμαστε σαφείς εδώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε και όλο το πρόβλημα της σύγκλησης των ε, κανονισμών και των ρυθμίσεων και η άποψή μας είναι ότι εξ αρχής Μια συμφωνία TTIP θα πρέπει να αποτελεί έναν κανονισμό αριστείας, εξαιρετικό εφόσον θα χρησιμεύσει αργότερα για άλλες διμερείς συμφωνίες. Έχουμε πράγματα τα οποία μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή, όπως το REACH, ε, στο οποίο επιμένουμε, είναι ένα σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των χημικών προϊόντων και δεν θα θέλαμε αυτός ο τομέας να αμφισβητηθεί από το TTIP πρέπει να εφαρμόσουμε τις κανόνες ε, εργασίας. Δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα, δεν είμαστε προστατευτικοί και επιμένουμε ώστε όλες οι χώρες να θέσουν σε εφαρμογή τους διεθνείς κανόνες που προτείνονται ή που θεσπίζονται από τον ε, Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Γνωρίζουμε ότι στη ΣΥΠΑ αυτοί οι κανόνες δεν έχουν επικυρωθεί, αλλά πιστεύουμε πως πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση και από αυτή την άποψη και το να πιστεύουμε πως ε, απλά παροτρύνσεις ε, για την εφαρμογή των κανόνων αυτών θα αρκέσουν δεν μας αρκεί. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ε, εμπορική συμφωνία με την Κορέα που παρά τις προσκλήσεις στα τρία τα συνδικαλιστικά δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά σε αυτή τη συμφωνία με την Κορέα. Ε, και κλείνω γιατί από ό,τι φαίνεται μακρυγόρησα, αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα θέματα, είναι αυξανόμενο ενδιαφέροντος για τους πολίτες αλλά και για τους τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους οποίους αντιπροσωπεύω ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ευρωεκλογών που σε λίγες εβδομάδε θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ γενναιόδωρος σήμερα. Λουίζα Σάντος, την έχουμε συνηθίσει να έρχεται εδώ. Εκπροσωπεί την Ένωση Κλωστεφαντουργικών ε, Προϊόντων και Ειδών Έντησης. Τώρα όμως είναι η κεφαλή του Διεθνούς ε, Τμήματος ε, της Διεθνής Διεύθυνσης από τη Business Europe. Συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που καλέσατε την ε, Business Europe ε, για να συζητήσει μαζί σας εδώ τα θέματα της ε, εμπορικής πολιτικής. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και θα περάσω στα βασικά. Και μετά βέβαια μεταχάς να ανεχθώ τις ερωτήσεις σας ως Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Business Europe γνωρίζουμε τι θέλουμε η εμπορική πολιτική να κάνει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τι μπορεί να κάνει. Όπως είπε και ο κύριος Αζεβέδο και η κυρία Ζεγκόλ, η εμπορική πολιτική δεν ε, εξασφαλίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Είπατε βιομηχανική πολιτική, κυρία Ζεγκόλ, εμείς συμφωνούμε από την Business Europe. Το επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να το δούμε με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για την εμπορική πολιτική, αλλά και άλλες πτυχές να αναφέρουμε, επίσης είναι σημαντικές και αυτές για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις και να συνεχίζουν να παράγουν στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Θέλουμε επίσης να δώσουμε ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, είτε για να εξαγάγουν εκτός Ευρώπης, είτε για να επενδύσουν εκτός Ευρώπης. Και εδώ ε, μπαίνει και το εμπορικό θεματολόγιο. Όπω και άλλοι ομιλητέ, και εμεί θα προτιμούσαμε την πολυμερή προσέγγιση. Φυσικά είναι η καλύτερη λύση ώστε συνολικά να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και στις αναπτυσσόμενες και στις ανεπτυγμένε χώρες. Τα προϊόντα δε, οι υπηρεσίες θα μπορούν να ρέουν και να κυκλοφορούν, ε, να κυκλοφορούν συγγνώμη, ελεύθερα μεταξύ των χωρών υπό αυτό το, με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε βέβαια σήμερα το πρωί ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό η Business Europe στηρίζει την πολυμερή προσέγγιση και δεσμεύεται στο πολυμερές θεματολόγιο στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα συναντηθούμε με τον κύριο Αζεβέδο σήμερα το μεσημέρι για να του πούμε ακριβώς αυτό, ότι θα στηρίξουμε δηλαδή ε, τον ΠΟΕ και τη δουλειά του κύριου Αζεβέδο για την προώθηση της ε, Ατζέντας. Πρέπει να είμαστε όμω και ρεαλιστέ. Οι επιχειρήσει χρειάζονται ευκαιρίε, συγκεκριμένε ευκαιρίε και αυτό και το διμερέ θεματολόγιο για μα αποτελεί μια εναλλακτική λύση που μάλιστα δίνει και κάποια αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι οι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου δεν είναι η μόνη εναλλακτική. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι για όσες χώρες δεν ε, υπάρχει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με αυτέ ή και αφού δεν υπάρχει ακόμη πολυμερή εμπορική συμφωνία, σε αυτέ τι περιπτώσει οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να εξάγουν, να παρέχουν υπηρεσίε και προϊόντα και στι ιδιωτικέ και στι δημόσιε αγορέ και να μπορούν να επενδύουν με του ίδιου όρου όπω και οι εγχώριε επιχειρήσει. Γι' αυτό ακριβώ η Business Europe θεωρεί ότι και η υλοποίηση των συμφωνιών, την Κορέα την αναφέραμε ήδη, αλλά και μια αποτελεσματική στρατηγική πρόσβαση στην αγορά. Σε αγορέ που δεν έχουμε συμφωνίε. δύο σημαντικές αναφέρθηκαν το πρωί, η Ινδία, δεν έχουν προχωρήσει πολύ ακόμη στις διαπραγματεύσεις και Μερκοσούρ. Βραζιλία κυρίως, πολύ σημαντική αγορά. Πρέπει να βρούμε λύσεις για τις αγορές αυτές, αλλά και για άλλες, όπως για τη Ρωσία, που και αυτή αναφέρθηκε σήμερα το πρωί. Πολυμερή θεματολόγιο, σύντομα, τι περιμένουμε από Business Europe. Περιμένουμε βέβαια το πακέτο του Μπαλί και ιδίω η συμφωνία περί διευκόλυνσης του εμπορίου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και εμείς ήμασταν στο Μπαλί ως Business Europe. Είμαστε ικανοποιημένοι με την έκβαση και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα περιμένουμε. Ε, θα τα γνωρίσουμε μόνο φέτος αυτά βέβαια, όταν οι χώρες θα κληθούν να πούν ποιες διατάξεις θα εφαρμόσουν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που περιμένουμε από τον ΠΟΕ είναι να ολοκληρωθεί δυνατόν ε, το θεματολόγιο της ε, Ντόχα. Αν όχι, θα πρέπει σίγουρα να διερευνήσουμε άλλα ενδεχόμενα. Ένα από αυτά είναι οι πολυμερείς συμφωνίες. Ο κ. Σαζεβέδο σήμερα το πρωί μίλησε για τη συμφωνία για τις υπηρεσίες, τη συμφωνία για τις τεχνολογίες που θα επεκταθεί, ίσως και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Ελπίζουμε και άλλες πτυχές που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο θεματολόγιο του ΠΟΕ να ανοίξουν στο μέλλον. Υπάρχουν και ακούστηκε και σήμερα από πολύ το θέμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων που είναι σημαντικό, αλλά και για μας είναι σημαντικό, παραδείγματος χάρη, το θέμα του ανταγωνισμού των επενδύσεων, των πρώτων υλών. Είναι πτυχές αυτές ε, τις οποίες συζητούμε και έχουν συζητηθεί και σε επίπεδο που ίσως να συζητηθούν εκ νέου στο μέλλον. Ο κ. Αζεβέδο έχει πολύπλοκο έργο και καθήκοντα σημαντικά να επιτελέσει. Ξέρουμε και βλέπουμε ότι είναι πολύ αποφασισμένος, δεσμευμένος να πετύχει ο ΠΟΕ κάτι και ο άλλος τομέας όπου θα μπορούσε να διαδραματίσει και θα έπρεπε να διαδραματίσει ρόλο που είναι στην ενσωμάτωση και ολοκλήρωση όλων των πολυμερών και διμερών συμφώνων που συνάπτονται. Δεν έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογή και Εύρο, είπε γι' αυτό τον μπολ με τα μακαρόνια, το σπαγκέτι μπολ ο κύριος Αζεβέδο. Πράγματι δεν είναι παντού τα ίδια, ούτε και το επίπεδο φιλοδοξιών είναι παντού το ίδιο. Νομίζω το Ποέ και εμεί από την πλευρά τη Business Europe πιστεύουμε ότι μπορεί ο ΠΟΕ να διδαματίσει και σε αυτό το ε, κομμάτι ε, ρόλο. Έρχομαι στη διμερή, στο διμερές θεματολόγιο. Δεν θέλω να εστιάσω υπερβολικά στη συμφωνία TTIP, διότι γνωρίζουμε ότι είναι μια συμφωνία ε, η κοινή γνώμη, ιδίως στην Ευρώπη, έχει αντιληφθεί τα πράγματα. Ε, έχουμε συζητήσει κατά πολύ το θέμα αυτό. Δεν είναι προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μόνο όμως η συμφωνία TTIP. Έχουμε τη συμφωνία με την Ιαπωνία, για παράδειγμα, που μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση, γιατί θα πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του τι έγινε μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων και έχουμε και τη συμφωνία ASEAN με το Βιετνάμ, με τη Μαλαισία, Ταϊλάνδη. Διαπραγματευόμαστε τις ε, διμερείς συμφωνίες με τις σημαντικές αυτές αγορές, ε, δυνητικά τουλάχιστον από πλευράς ανάπτυξης και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε θετικά και μια σημαντική συμφωνία με τον Καναδά συγκεκριμένα. Συνεχίζει λοιπόν το διμερές ε, μέτωπο να έχει άλλες σημαντικές προτεραιότητες για την Business Europe. Αλλά θα πρέπει να σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι το TTIP είναι παρελθόν ένα προτεραιότητα για εμάς ό,τι αφορά τις μερικές συμφωνίες. Για ποιο λόγο. Διότι έχουμε ολοκληρωμένε οικονομίε, ε, είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επαναλάβω πόσο σημαντικέ είναι οι μεταξύ μα σχέσει. Είναι πραγματικότητα όμω σήμερα. Και πιστεύουμε ότι λαμβάνοντα υπόψη τα μεγέθη των οικονομιών και το επίπεδο ανάπτυξης, μια τέτοια συμφωνία δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει ωφέλη και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Το πιστεύουμε αυτό διότι αντίθετα με όσα ισχυρίζονται ορισμένοι, δεν θα μειωθούν τα πρότυπα σε πολλούς τομείς. Τι εννοώ, για παράδειγμα, το ρυθμιστικό σκέλος το έθεσε και προλαλήσασα. Δεν θέλουμε μείωση ε, του επίπεδου των ε, προτύπων για τις περιβαλλοντικές πτυχές ή το ρίτς για παράδειγμα ε, σε σχέση με αυτά τα πρότυπα. Θέλουμε όμως ορισμένοι κανονισμοί που συνιστούν αλληλεπικάλυψη να συγκλίνουν τουλάχιστον μεταξύ τους ή να καταργηθούν αυτές οι αλληλεπικάλυψεις. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Καλλιντικά υπάρχει ενημέρωση της, ε, για τη σύνθεση των προϊόντων. Το νερό που είναι ένα συστατικό των προϊόντων αυτών, θεωρητικά θα πρέπει να μεταφράζεται στις διάφορες γλώσσες. Όμως, οι επιχειρήσει ε, συμφώνησαν και υπάρχει διεθνέ πρότυπο που λέει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λατινική λέξη άκουα για να ορίζουμε το νερό. Αυτό είναι παντού αποδεκτό πλην στη ΣΥΠΑ, όπου απαιτείται να μπαίνουν και τα δύο. Aqua και water στα αγγλικά, το νερό. Εμείς θέλαμε να ε, αποφύγουμε κάθε φορά που στέλνουμε ένα προϊόν στις ΙΠΑ να ε, πρέπει να αλλάζουμε τις συσκευάσεις και να βάζουμε και τη λέξη νερό. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα κλωστοϊφαντουργικά. Στις ετικέτες έχουμε, ξέρετε, όλα αυτά τα σύμβολα για το πώς πλένονται τα ρούχα κτλ. Αυτά τα σύμβολα είναι σχεδόν, τα ίδια, σχεδόν παντού τα ίδια. Ή είπα, έχουν και εκεί διαφορέ. Και εμεί αυτό που θέλουμε κατά βάση είναι να δεχτούν τα δικά μα σύμβολα, γιατί οι διαφορέ είναι ελάχιστε, είναι πολύ μικρέ. Και δεν είναι πρόβλημα του καταναλωτέ αυτό, Αντιθέτω. Θέλουμε οι εταιρείε να αποφύγουν κάθε φορά που εξάγουμε ή θέλουμε να εξάγουμε στι αγορές να πρέπει να φτιάξουμε διαφορετική ετικέτα. Αυτά είναι δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα ε, του πώ. Ε, μια συμφωνία ε, σαν το TTIP μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Και έρχομαι και στους καταναλωτές, οπότε μπορεί να βοηθήσει και τους καταναλωτές. Για ποιο λόγο. Διότι ακόμη και αν από πλευράς δασμών είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχετικά χαμηλούς δασμούς, έχουν στα ε, προϊόντα υψηλούς δασμούς, της τάξης του 20 έως 30% ορισμένες φορές. Μια ε, μικρομεσαία επιχείρηση στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία που θέλει να εξαγάγει ε, ένα τελικό ε, προϊόν στις Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να πληρώσει 20% δασμό. Και παρότι εμεί δεν έχουμε τόσο υψηλό δασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάποια γεωρικά προϊόντα ναι, αλλά όχι στα βιομηχανικά αγαθά τόσο, πάντως αυτό κάνει τη διαφορά. Αν δηλαδή ένας καταναλωτής θέλει να αγοράσει ένα προϊόν made in USA, είναι διαφορετική η τιμή που θα πρέπει να πληρώσει αν έχει να καταβάλει 10% δασμό. Αυτό θα μετακυληθεί στην τελική τιμή. Αν είναι μηδενικό ο δασμό, σίγουρα θα είναι φθηνότερο το προϊόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτά λοιπόν τα συγκεκριμένα παραδείγματα ε, δείχνουν πώ μπορεί να ωφελήσει αυτή η συμφωνία. Και επίση μπορεί να ωφελήσει και του εργαζομένου. Όπω προείπα, δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία. Εγγύηση όχι, δεν αποτελεί. Όμω, αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περισσότερε ευκαιρίε να κάνουν εξαγωγέ. και σα εξήγησα πώ. Αν αναπτύξουν περισσότερο την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είναι φυσιολογικό να επενδύσουν περισσότερο και άρα να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Θα ε, σταματήσω εδώ σε διαφορά τη συμφωνία TTIP και θα κλείσω με ένα σημείο που είναι σημαντικό για εμάς και για εμάς. Έχει ήδη αναφερθεί. Πολλοί το είπαν και οι προλαλήσασα. Είπαμε ότι το ελεύθερο εμπόριο δεν θα πρέπει να φτάσει στα άκρα Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε και για την, τον εξεχρονισμό του μηχανισμού και των μέσων εμπορική άμυνα. Εμεί, στην Business Europe ε, στηρίζουμε πάρα πολύ και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτόν τον εξυγχρονισμό και ελπίζουμε να πετύχει απτά αποτελέσματα αυτή η διαδικασία. Βεβαίω και μας ανησυχεί το επίπεδο των διαφόρων που υπάρχουν μεταξύ της θέσης του Συμβουλίου και της θέση του Κοινοβουλίου. Όμως ελπίζουμε ότι τελικά θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία εξυγχρονισμού. Πρέπει να σας πω όμως ότι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι σημαντικό να βρεθεί συμβιβασμός. Αμφότερες πλευρές πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς σε σχέση με τη θέση που έχουν υποβάλει. Δεν θα συζητήσω το κοινωνικό ντάμπινγκ, το οικονομικό ντάμπινγκ. Θέλω να σας πω απλά ότι έχουμε τους κανόνες του ΠΟΕ και πρέπει να τους στηρίσουμε, τους κανόνες αυτούς. Αυτό το εργαλείο είναι οικονομικό. Δεν πρέπει να το ε, πολιτικοποιήσουμε σε υπερβολικό βαθμό. Πρέπει να λειτουργεί σε οικονομική βάση. Και είναι σημαντικό να λειτουργεί. Και ελπίζω και με αυτό ολοκληρώνω ότι και οι δύο πλευρές θα επιδείξουν κοινή λογική, κοινό νου για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, κάτι που είναι σημαντικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιχειρήσεις εκείνες που θέλουν να εισαγάγουν προϊόντα ή να τα χρησιμοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, παράγουν αγαθά μεγαλύτερη προστέμενη αξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σταματώ εδώ και περιμένω τις ερωτήσεις. Thank you both of you. Uh, the floor is open for the members of this. Uh... Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ, όποιος θέλει το λόγο. Bernd Lange was the first one. SND, floor is yours. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal... Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στο ερώτημα της, της τεκμηρίωσης των κοινωνικών και τεχνολογικών προτύπων. Τα όσα είπε η οργάνωση, η συνομοσπονδία δηλαδή των ε, οργανώσεων εργατικών συνδικάτων μίλησε για ένα gold standard εκπρόσωπός τους που θα πρέπει να θεσπιστεί. Διερωτώ αν και η Business Europe δεν θα έπρεπε να κινηθεί προς παρόμοια κατεύθυνση βλέποντας και τις πολλές προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλιστεί μια άσκηση επιρροής και προς άλλους εταίρους. Και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πρότυπα και σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ώστε να θεσπιστούν κάποιες λογικές ρυθμίσεις και με την έννοια αυτή νομίζω δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς κάπως αφελώς ότι οι αρκούν οι εμπορικές σχέσεις για να εξασφαλιστούν οι καλές συνθήκες εργασίας. Με άλλα λόγια, δέχεστε απλά το dumping που ενδέχεται να προέλθει από ορισμένες ρυθμίσεις. Sturdy για την Business Europe. δεν μιλήσατε για την Europe Career, για την εφαρμογή και για την ISTS, για τη συμμετοχή της στην ΣΥΤΑ, της Σιγκαπούρης, καθώς και τις άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών για το μέλλον. Κατρίν Βιέρντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και τόσο γρήγορα κιόλας. Έχουν ήδη ακούσει παρόμοιες ερωτήσεις από μένα οι συνάδελφοί μου και ίσως είναι κάπως στενή η ερώτησή μου. Προέρχομαι από το Ενωμένο Βασίλειο και θα γνωρίσετε τη συζήτηση που γίνεται στο Ενωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο επηρεάζει το εμπόριο. Και το να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι συμμετέχει και ως μέλος ενός μπλοκ στη διαπραγματεύσεις για το εμπόριο. Και για το αν θα αποφασίσει τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο, αν θα μείνει ή αν θα φύγει, θα λέγατε εσείς ότι είναι πλεονέκτημα για τους πολίτες της Ένωσης να μπορούν να διαπραγματεύονται ως μέλη ενός συνόλου, αλλά και για την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι πλεονέκτημα ή θα προκύψουν σημαντικά μειονεκτήματα εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σόλτς από την Ενωτική Αριστερά. Πολύ σημαντικό που παρίσταστε εδώ. Μετά από τα όσα ακούσαμε και από τον Γενικό Διευθυντή κύριο Αζεβέντο για τα πολυμερή συστήματα. Η κυρία Σεγκόλ είπε ότι μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στο εμπόριο, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Μιλήσατε και για την συμφωνία με τις ΗΠΑ. Έχετε όμως φτιάξει και μια ομάδα εργασία. Ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που βλέπετε και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενοποίηση των προτύπων και πώς μπορεί να εφαρμοστεί και από τους δύο εταίρους. Και αυτή είναι ερώτηση και προς την Business Europe. Χθες ακούσαμε για τη μελέτη του ρυθμιστικού μηχανισμού και πώς συνδέει τις νομοθετικές διαδικασίες και τους κανονισμούς οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να προκύψουν και βέβαια τις ξεχωριστές ρυθμίσεις που κάνουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η θέση της Business Europe για αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πού βλέπετε να βρίσκεται ο ρόλος σας και η ευθύνη σας. Να συμμετάσχετε δηλαδή στην προσπάθεια δημιουργίας απασχόλησης. Και θεωρείτε ότι η μελέτη αντικτύπου μπορεί να σημάνει ότι θα δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το πιστεύετε αυτό ή θεωρείτε ότι μάλλον είναι συνοδευτικό, συνοδευτική η επίπτωση αυτή των ρυθμίσεων αυτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, εσείς. Dartmouth. Είπε η κυρία Μπίαντερ ότι διεξάγεται μεγάλη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για το εάν θα πρέπει να παραμείνει η χώρα αυτή στην ε, Ενωμένη Ευρώπη ή όχι. Και έχει ορισμένες ερωτήσεις. Έχω καλά νέα, Κάθριν. Επιτέλους, ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές σου. Στις τελευταίες συνεδριάσεις είπα ότι φτιάχνω, γράφω ένα βιβλίο και λέω να φύγουμε από την Ένωση να βγούμε στον κόσμο. Έχω φτάσει στις 30.000 λέξεις και το έχω στείλει στο τυπογραφείο. Ό,τι ήθελες να μάθεις πάντοτε αλλά φοβόσου να ρωτήσεις τα βάζω όλα εκεί. Ξαναλέω, οι προσευχές σου εισακούστηκαν και θα στείλω αντίγραφα και στα άλλα μέλη της Επιτροπής αλλά και στη Γραμματεία. Αναγνώριση για τις προσπάθειες του κυρίου Μορέιρα και για το ότι όσα έχουν κάνει ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια να μου βοηθήσουν να κατανοήσω την, ουσία του θέματος. Ε, ε ευχαρίστως, να, φύγετε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, λέει ο πρόεδρος. Τώρα να έρθω σε αυτά που είπε η κυρία Σεγκόλ. Αφού συγχαρώ πρώτα την κυρία για το εύγλωτο των της ομιλίας της, ακόμα και μέσα από τη μετάφραση. Αν ήξερα γαλλικά θα είχα μείνει έκθαμβος. Λίγα σχόλια τώρα, πολύ σύντομα και έχω δύο ερωτήσεις. Συμφώνησα με την κυρία Σεγκόλ για τη διαφάνεια. Εμείς είμαστε λίγαν υπέρ της διαφάνειας Πάντα υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας της ενωτικής αριστεράς όταν ζητούν διαφάνεια για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, υποστηρίζουμε την οργάνωσή σας όταν απαιτεί τη διαφάνεια. Όμως, εκτός από αυτό δεν νομίζω να συμφωνώ σε πολλά άλλα. Εσείς μιλείτε για βιομηχανική πολιτική, μα δεν έχει και πολύ σχέση με τις αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής Εμπορίου η βιομηχανική πολιτική έχει απολέσει την αξιοπιστία της στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα και δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει, διότι οι αξιωματούχοι των διοικήσεων δεν λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Ούτε όταν εμείς το, το επιδιώξαμε, ούτε όταν η Γαλλία προσπάθησε, δεν, επέδωσε, δεν απέδωσε η προσπάθεια αυτή. Μιλήσατε ακόμη για την κοινωνική διάσταση που περιλαμβάνεται και σε μια από τις συνθήκες. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Ίσως μπορείτε στις απαντήσεις σας να μου πείτε σε ποιο άρθρο, ποια συνθήκης περιλαμβάνεται αυτό. Δεν θελήσατε να μιλήσατε στα αγγλικά, αλλά εγώ θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μου το εξηγήσετε. Ίσως υπάρχει όμως μια ασυμβατότητα μεταξύ της επιβολής μιας κοινωνικής διάστασης και της επίτευξης οικονομικής ευημερίας και απασχόλησης. Για παράδειγμα, έχουμε όλες αυτές τις πράσινες πολιτικές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρη λόγω αυτών έχουμε πολύ ακριβότερες τιμές ενέργειας, περίπου δύο ή τρεις φορές περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μία από τις ηρωνίες αυτές είναι ότι βεβαίως τα συνδικάτα θέλουν να διατηρηθεί η χαλιβουργία και ούτω, καθε, και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά είναι αντιφατικά. Και όπως είπε η κυρία Σάντος, ο πρόεδρος, μπορείτε να βάλετε τις ερωτήσεις σας, να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Υπάρχουν κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά αυτό που προτείνεται είναι μια πρόσθετη διάσταση που να έρθει σαν καπάκι από πάνω. Και έχω τέλος και μια ερώτηση για την κυρία Σεγκόλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Στο άρθρο 6. Βλέπετε εσείς να υπάρχει καμιά ασυμβατότητα οποιαδήποτε κατά την άποψή σας μεταξύ υψηλών μισθών και ελεύθερης διακίνησης εργατικού δυναμικού από πολύ, χαμηλέ, από ε, πτωχές χώρες. Διότι γνωρίζουμε ότι τελικά το κατακεφαλήν εισόδημα του Ηνωμένου Βασιλείου μειώνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία διόρθωση. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης εδώ και 10 χρόνια περιλαμβάνουν ρήτρα για τα δικαιώματα εργασίας και όλες οι αμερικανικές από την αύτα και μετά εδώ και 20 χρόνια δηλαδή όλες περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εξαναγκαστικές ρήτρε για τα δικαιώματα των ε, εργαζόμενων. Ναι, ναι, βεβαίω, είμαι βέβαιος, αλλά δεν απαντάτε με αυτό στις ερωτήσεις μου. Ρωτήσατε πού είναι, ε, λέει ο πού είναι. όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν ερώτησα ε, αυτό. 20 δευτερόλεπτα δώστε μου. Παρακάλεσα η κυρία Σεγκόλ που διάβασε ένα από τα άρθρα από κάποιες από τις συνθήκες της Ένωσης. Όχι, δεν προσπαθούσα να κάνω κάποια παραπλανητική ερώτηση. Ήθελα να μάθω ποιο άρθρο από ποια συνθήκη. Το υπαριθμό 21 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρφυ. Ε, γίνονται εκλογέ στη Βρετανία, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Δύο ερωτήσει τώρα προς την κυρία Σεγκόλ. Πρώτα γενική ερώτηση για τη σημασία της εμπορική πολιτικής από την άποψη των εργατικών συνδικάτων. Μου φαίνεται ότι είναι και όλο και πιο σημαντικό θέμα. Όχι, δεν είναι μόνο ζήτημα αλληλεγγύης με τους αδελφούς μας άλλων χωρών που συμμετέχουν σε εμπορικές συμφωνίες, ούτε μόνο για θέμα dumping πρόκειται. Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία του κατεστημένου των ε, επιχειρήσεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ε, επιχειρηματική πολιτική σαν ε, δούριο ύπο για να υπονομεύσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί καθαρά από το εργατικό κίνημα. Και σε ό,τι αφορά την ρυθμιστική σύγκριση, συγγνώμη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρόκειται μοναχά για aqua, water και διάφορα τέτοια στα καλλιτικά. Πιο πολύ είναι το θέμα του STS, και των συμφωνιών ΣΥΤΑ που ανοίγουν ολόκληρη, ολόκληρο αριθμό υποθέσεων κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Τέλος, ακούσαμε πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως για την εποχή μετά την άκτα για διαφάνεια συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών κλπ. Άλλαξε τίποτα. Υπάρχει πραγματική ίση συμμετοχή για σας όπως υπάρχει για την Business Europe ή άλλες οργανώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Merci, Monsieur le Président. Euh, deux petites questions. Euh, une première. Ζαντώ, δύο σύντομες ερωτήσεις προς την κυρία Σεγκόλ με τον ένα τον άλλο τρόπο συμμετέχετε, έχετε κάποια σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο, το με ανάπτυξη των διαπραγματεύσεων με το Καναδά. Γιατί μας δόθηκε να καταλάβουμε ότι ναι, είναι πολύ ικανοποιημένος ο κ. Μπαρόσο που ανακοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη τίποτε, Ιδίω στο κοινωνικό κεφάλαιο και για την κυρία Σάντος ένα ερώτημα. Θεωρείτε ότι είναι καλό νέο το γεγονός ότι δυνητικά η Κομισιόν θα εγκρίνει ένα νέο γενετικό τροποποιημένο αραβόσιτο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με, τον, με που το αναφέρω αυτό. Πρόεδρος, ε, ο κύριος ε, Μικελάντζελο ή κάπως έτσι από την Κομισιόν θέλει το λόγο, όχι. Να δώσω τώρα το λόγο στις κυρίες, αλλά θα ξεκινήσω ανάποδα. Δηλαδή θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Σάντος. Μάλιστα. αφήστε να πω εγώ τα δικά μου και μετά αν έχω ξεχάσει κάτι με διορθώνετε. Κύριος Λάγκε, κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Νομίζω ότι στην Business Europe Είχαμε έρθει εδώ στην Επιτροπή σας και κατά το παρελθόν για να συζητήσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, στηρίζουμε τη συμπερίληψη του κεφαλαίου της βιωσιμότητας ε, στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και όπως νομίζω ότι προανέφερα στην πρώτη μου παρέμβαση, αυτό το θέμα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο θεματολόγιο του ΠΟΕ. Και ήταν και στο θεματολόγιο τη Σιγκαπούρη, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο. Μέρο των όσων πρέπει να γίνουν θα εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη τη κυβερνήση και ένα άλλο από τι επιχειρήσει. Τώρα, από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι ξεκάθαρο ότι πολλέ από τι επιχειρήσει μα, επειδή έχουν παγκοσμιοποιημένε αλυσίδε ε, εφοδιασμού που δύσκολα κανεί μπορεί να ελέγχει ε, ορισμένε φορέ. Υπάρχει πολιτικές ε, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, τις οποίες εφαρμόζουν περισσότερες επιχειρήσεις και ιδίως αυτές που ε, δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν ε, υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας σε παγκόσμιο Και αυτό το στηρίζουμε. Αυτό που δεν θέλουμε και νομίζω ότι αυτή είναι η θέση μας προς το παρόν, δεν θέλουμε οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου να χάσουν το βασικό στόχο που έχουν. Ότι είναι δηλαδή μια συμφωνία, είναι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, απελευθέρωση του εμπορίου. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος ο στόχος. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αυτό που μπορεί να συμβεί, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ινδίας, και με κάποιε άλλε από τι χώρε που διαπραγματευόμαστε είναι ότι δεν θέλουν ορισμένε χώρε να μπει αυτό το κεφάλαιο στι συμφωνίε ελευθερών εμπορίου όπω είδαμε ξεκαθαρά με την Ινδία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε σήμερα για δημιουργία αποδομών, ικανοτήτων, πώ μπορούμε να επηρεάσουμε τι χώρε να αλλάξουν ε, άποψη. Όμω δεν μπορούμε να του υπαγορεύσουμε τι πρέπει δεν πρέπει να κάνουν, να τι ενθαρρύνουμε, να τι παρακινήσουμε, να κάνουν περισσότερα μπορούμε. Υπάρχει όμω και ένα όριο στο τι μπορούμε εμεί να κάνουμε. Και νομίζω ότι ο κύριος Ασεβέδο το πρωί, απαντώντας σε ορισμένα ερωτήματα, το ξεκαθάρισε. Είναι καλύτερα, μάλλον σημαντικό να συνεργαστεί καλύτερα ο ΠΟΕ με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος οργανισμός σε πολυμερές επίπεδο που να συνδυάζει τις τρεις πτυχές που επηρεάζουν το ε, εμπόριο κυρίως, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ίσως. Φυσικά και δεν είμαστε όμως κατά της αηφόρειας, κατά της βιωσιμότητας. Σε καμία περίπτωση. Για τον κύριο Στέρντι. Κορέα. Εφαρμογή, εφαρμογή ελεύθερων, συμφωνίων ελεύθερου εμπορίου. Όπως προανέφερε είναι μια από τις ε, διαστάσεις που πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει, να δοθεί έμφαση, όπως και από πλευράς Κομισιόν, διότι είμαστε στην τελική φάση ε, με, για ορισμένες συμφωνίες και δεν και κάποιες άλλες. Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της υλοποίηση, που θα προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Μίλησα για την γενική στρατηγική πρόταση στις αγορές. Εννοούσα και το σκέλος εδώ της εφαρμογής, γιατί και πάλι σήμερα το πρωί ο κύριος Ζαβέδο πρέσβη τον λέω, τέλος πάντων, ο κύριος Σαζεβέδο ανέφερε το ρίσκο οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες να οδηγήσουν σε αύξηση των μέτρων των προστατευτικών στον τομέα ιδίω στο ρυθμιστικό, στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει, δεν αρκεί η συμφωνία, να φροντίσουμε μετά τη συμφωνία να δούμε τι γίνεται στο, με την εφαρμογή. Με την, Κορέα το είδαμε. Και είναι σημαντικό και στην επιθετική στρατηγική της Ένωσης, ε, συμπληρωματικά προς την πολιτική με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Για το ESTS, επειδή ετέθησαν και άλλα ερωτήματα. Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει την επίσημη θέση μας. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε υπέρ του να συμπεριληφθεί σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερο να για τη Σιγκαπούρη, για τον Καναδά, για τις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι η συμπερίληψη της διάστασης αυτής δεν θα οδηγήσει σε ανάλαφους ισχυρισμού και αξιώσεις από επιχειρήσεις ε, αμερικανικές που θα επηρεάσουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, γιατί δεν το πιστεύουμε, δεν θέλω να σας το αναλύσω, αν θέλετε μπορώ. Αλλά ως επιχειρήσεις είμαστε ανοιχτοί στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης για να διασκεδαστούν μέσα από τις ανησυχίες που ετέθησα. Θεμητές ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, κάποιες οφείλονται και στην έλλειψη ενημέρωσης για το τι ακριβώς είναι το ESTS, πώς μεταφράζεται Πρέπει να έχουμε μια επικοδομητική προσέγγιση, θεωρούμε όμως ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η διάταξη αυτή, γιατί δεν αξιοποιούμε ή δεν αξιοποιείται, μάλλον δεν χρησιμοποιείται ή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι αλαφρά τη καρδία αυτό το εργαλείο. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει να χρησιμοποιείται τα κτλ. Το θέμα είναι όταν αλλάζει άρδινο ένα σύστημα, όχι για, μικρά, για μικρές σαλή. Όταν αλλάζει άρδινο ένα σύστημα θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα μια εταιρεία να προσπαθήσει μέσω ενός ανεξάρτητου συστήματος να επιλύσει αυτά το προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι σύντομη, αλλά τι να κάνω. για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κύριο Μέρφυ έφυγε, γι' αυτό θα μιλήσω. Τέλος πάντων, για το ρυθμιστικό σκέλος όμω. Φυσικά και θέλουμε σύγκληση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε και το επίπεδο των προτύπων ή το επίπεδο της προστασίας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο. Επίσης πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα θέσει ένα γενικό πλαίσιο μεγάλο μέρος της δουλειάς που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει από, τις, ε, από τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις προς τους διαπραγματευτές για το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα συγκεκριμένα προβλήματα που υφίστανται. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη ρυθμιστική συνεργασία και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Πρόεδρος. Έχετε μισό λεπτό. Ah, Frankly, uh, considering... Η απόφαση βγήκε χτες. Σε σχέση με τις αποφάσεις ε, για το ESTP ε, ε, και τις άλλες, δεν βλέπω να έχουν αυτές αντίκτυπο. Αυτό που βλέπω να έχει αντίκτυπο είναι αυτό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συναντηθούν ο πρέσβης Φρόμ και ο επίτροπος Τιγκούχτ, ώστε να κάνουν μία αποτίμηση της κατάστασης και δεύτερον, ώστε να ε, ε, φτιάξουν ένα πολύ φιλόδοξο ε, χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και το λόγο έχει η κυρία Σεγκόλ. Εγώ θα είμαι σύντομη. Είχα όμως τρεις ερωτήσεις από Βρετανούς συναδέλφους Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για Βρετανο-Βρετανική συζήτηση. Ναι, βεβαίω, αλλά χρησιμοποιώ τα αγγλικά για να είμαι βέβαιο, βεβαία ότι καταλάβατε πώ ξέρω αγγλικά. Ναι, βεβαίω. Είμαστε ισχυρότεροι εφόσον διαπραγματευόμαστε από κοινού. Και αυτή είναι η σύντομη μου απάντηση σε μια σύντομη ερώτηση. Η διαφάνεια είναι βεβαίως, βεβαίως ναι. Αλλά θέλω να θυμίσω εδώ ότι αυτό που έχουμε ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα κοινωνίας και δεν είναι απλά, δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αφορά ένα συγκεκριμένο είδος κοινωνίας. Το να λέμε λοιπόν ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να αποκλείεται για μας σημαίνει το τέλος αυτού του οράματος. Εφόσον δεν υπάρχει κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι πολίτες και οι ψηφοφόροι και οι εργαζόμενοι δεν είναι, θα είναι σε θέση να ξεκολουθήσουν να το στηρίζουν. Και η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητη, απολύτως απαραίτητη. Δεν μίλησα για ψηλά ημερομίσια. Είμαστε υπέρ τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπω είναι αυτή θεσπισμένη και με τα όρια που υπάρχουν στην Ένωση για όλου του εργαζόμενου, από οποιαδήποτε η προέλευσή του, η εθνικότητά του και το ημερομίσθιό του και ο μισθό του. Ο κύριο Μέρφυ έχει φύγει, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποιο θα του μεταφέρει την... τι πιστεύω για το Άλλο, για τον Δούριο ύπο, Ναι, θέλουμε διαβουλεύσεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν είναι απαραίτητος δούριο Ήπος, αλλά δυνητικά. Και σίγουρα στην συμφωνία ΣΥΤΑ δεν συμμετείχαμε επαρκώς και είναι αλήθεια ότι η ρυθμιστική σύγκληση θα μπορούσε να εξαλειχθεί σε απορρίθμιση και αυτό δεν το επιθυμούμε. Οπότε θέλουμε να συμμετέχουμε μόνο και μόνο για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πατήσω στο, στα γαλλικά στον κύριο Σόλτ. Δυστυχώ τα γερμανικά μου δεν με βοηθούν. Όντως έχουμε επαφές και συζητήσεις με τα αμερικανικά συνδικάτα και τα σημεία που προέταξα, είτε πρόκειται για τη διαφάνεια, είτε πρόκειται για τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι σημεία τα οποία συμμεριζόμαστε. Και θα έλεγα ότι από πλευράς της FACIO υπάρχει επιθυμία διάφορα συνδικαλιστικά δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα ιδιαίτερα για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την κατάρτιση να μεταφραστούν σε συμφωνίες όπως ε, αυτές αυτού του είδους. Ολοκληρώνω, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι μακρηγόρησα στην απάντησή μου. Ε, και για τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, όχι. Δεν συμμετείχαμε. Δεν γνωρίζω το κείμενο της συμφωνίας. Και δεν ε, μπόρεσα να δεις στα συρτάρια της Business Europe για να δω αν έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Αλλά πάντως εμείς δεν, δεν ε, μπήκαμε μέσα στα άδυτα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, τώρα ολοκληρώνεται η δημόσια μας συνεδρίαση. Θα έχουμε τώρα συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών με τους συντονιστές. Παρακαλώ τους συντονιστές μόνο λοιπόν να παραμένουν και οι υπόλοιποι να εγκαταλείψετε την αίθουσα γιατί έχουμε πάρα πάρα πάρα πολύ αργήσει στο πρόγραμμά μας.